Θα δώσω το λόγο εκ μέρου του Συμβουλίου στον κύριο Νταϊλαβέντοβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Συμβουλίου να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία και να σας συγχαρώ για το βραβείο Καρλομάγνο που παραλάβατε. Στην σύνοδο του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, δύο θα είναι τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα των επενδύσεων και αυτό της Ουκρανίας. Η χρηματοπιστωτική κρίση, η κρίση του χρέους, έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη θέση να ξανασχεδιάσει την οικονομική της στρατηγική. Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βρίσκεται στο κέντρο αυτής της στρατηγικής, όπως και οι επενδύσεις. Θα βρεθούν στο κέντρο της προσοχής του Συμβουλίου. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από επενδύσεις. Υπάρχει βεβαίως ένα τεράστιο αποθεματικό προγραμμάτων αξιοσημείωτο αποθεματικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, αλλά τα φιλόδοξα προγράμματα δεν είχαν πάντοτε των κατάλληλων επενδύσεων, ακόμη και όταν οι δυνατότητέ του σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τεράστιε. Προφανώ υπάρχουν λόγοι για την κατάσταση αυτή και η κρίση είχε έναν πολύ σοβαρό αντίκτυπο στη συμπεριφορά όλων των κρατικών, οικονομικών ε, φορέων και των ιδιωτών επενδυτών. Η επιφυλακτική τους στάση, λόγω της αβεβαιότητας για το κέρδος, ε, έχει εμποδίσει την, ε, την πρόοδο. Αλλά αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Ένας από τους βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι λοιπόν να ε, τονώσει την εμπιστοσύνη. Πρέπει να έχουμε περισσότερες επενδύσεις και να βελτιώσουμε το επενδυτικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δώσει προσανατολισμούς και κατευθυντήριες γραμμές για τους βασικούς επενδυτές σε πρώτη φάση μεταξύ του θεσμού ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Στατικές Επενδύσεις ε, που θα αναλάβει τη λειτουργία, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του μεταξύ του 2015 και 2016, εκεί θα χρειαστεί η κοινή στήριξη των δύο θεσμικών οργάνων. Ω συνομοθέτε, θα πρέπει πολύ γρήγορα να λάβουμε μέτρα για την νέα νομοθετική πρόταση, ώστε οι νέε επενδύσει να ξεκινήσουν αμέσω, στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να ε, συνδράμει αυτές τις δραστηριότητες με δικούς της πόρους. Σε δεύτερη φάση, με τη συνέχιση των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και την εξυγίανση των κρατικών δημοσιονομικών, θα πρέπει να ευνοηθεί η ανάπτυξη. Αυτέ είναι οι βασικέ προποθέσει για την ανάπτυξη. Δεν μπορούν να υπάρξουν επενδύσει εάν δεν είναι υγιή τα δημοσιονομικά του κάθε κράτου, με δημοσιονομική σταθερότητα και νομοθετική βεβαιότητα με, τα, με την δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που να είναι προβλέψιμο για τις επενδύσεις, ο ρόλος μας ως συνομοθετών θα είναι καθοριστικός. Προκειμένου να βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να ε, έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προκειμένου να βελτιωθεί και η νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο θα ε, εκφράσει πολιτικούς προσανατολισμούς και θα καταρτήσει και προτεραιότητε ανάλογα με τι αρμοδιότητε και τι ευθύνε του όπω ορίζονται στι συνθήκε. Τώρα, το να μεταφραστούν αυτοί οι προσανατολισμοί και προτεραιότητε σε πραγματική οικονομία είναι η βασική δική μα αρμοδιότητα. Η δική μα ευθύνη. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ε, αναλάβουν δράση άμεσα και εντατικά για να φανούν στην πράξη κατά αποτελέσματα που περιμένουν από εμά οι πολίτε μα. Ε, το Συμβούλιο, και μπορώ να μιλήσω και εκ μέρου τη Λετωνία που θα διαδεχθεί την Ιταλική Προεδρία, θα κάνει ό,τι μπορεί για να καταρτήσει αυτό το πλαίσιο για τι επενδύσει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είστε εξίσου αφοσιωμένοι στον ίδιο στόχο με εμά, όπω φάνηκε και πριν από λίγε εβδομάδε κατά τη συζήτηση για το επενδυτικό πρόγραμμα για την Ευρώπη, όπω προτάθηκε από τον πρόεδρο Γιούνκερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με έναν σύντομο σχόλιο για την Ουκρανία, όπου η κατάσταση παραμένει αρκετά επισφαλής. Οι εξελίξεις στα ανατολικά της χώρας είναι πηγή βαθιών ανησυχιών. Ε, ξέρουμε ότι τέτοιες ανησυχίες είναι ανησυχίες που αποσχολούν και πολλού πολλούς βουλευτές. Οπότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθήσει στενά το τι μπορεί να γίνει για τι εξελίξει αυτέ και θα δει κατά πόσο μπορεί να αναλυθούν νέε πρωτοβουλίε εφόσον χρειάζεται. Όπω ξέρετε, αυτή την εβδομάδα η είπατε πρόσωπο ε, Φεντερίκα Μογκερίνη βρέθηκε στο Κίεβο και θα ε, ανακοινώσει στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα τη επίσκεψή τη. Η κατάσταση στην Ουκρανία ε, απαιτεί από την νέα κυβέρνηση να εφαρμόσει νέε βαθιέ μεταρρυθμίσει. Θα πρέπει να του ενθαρρύνουμε και να του στηρίξουμε στην προσπάθειά του προκειμένου να αναμορφωθεί γενικότερα η χώρα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και περιμένω τι ε, παρατηρήσει και τα σχόλιά σα. Το διαβεβαιώνω θα μεταφερθούν στον πρόεδρο Τούσκ πριν από την αυριανή σύνοδο. Άλλωστε, ο πρόεδρος θα συμμετάσχει και στην ολομέλειά σας του Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστώ κύριε Νταλαβέντοβα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρόεδρος Γιούνκα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που έχω δυνατότητα να σας παρουσιάσω την άποψη της ε, Επιτροπής για την συνάντηση κορυφής και θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να μεταδώσετε, να μεταβιβάσετε την άποψή μου στους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι είναι καλό να, να ενημερωθούν. Οι συνάδελφοι ε, είναι καθοδόν κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ο Πρόεδρος Σούλς για να μεταβάσουν στο εκλογικό του σώμα το μήνυμα που αποστήλατε χθες. Προσβλέπουμε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα θα συζητηθεί η νέα προσέγγιση για τις επενδύσεις και πρέπει να επικεντρωθούμε στην βελτίωση της επενδυτικής ατμόσφαιρας που επικρατεί στην Ευρώπη. Πρέπει να βοηθήσουμε επίσης την ανατολική γειτονά μας, την Ουκρανία, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του χειμώνα και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην επιτυχή εφαρμογή των στόχων μας. Θα αρχίσω με κάποιες παρατηρήσεις για τη νέα μα αυτή προσέγγιση όσον αφορά τις επενδύσεις. Στις 28 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το... την έρευνά της που αναφέρεται στην απασχόληση και στο επενδυτικό πακέτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσήγηση που βασίζεται σε διάφορους πυλώνες που πρέπει όλοι μαζί να εφαρμοστούν και να συνεργαστούμε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι χώρες μέλη προκειμένου να πετύχουμε αποτελέσματα από τα οποία να επωφεληθούμε μακροπρόθεσμα. Επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις, προώθηση της δημοσιονομικής ευθύνης, υπεύθυνη επίσης ε, συμπεριφορά όσον αφορά την ε, ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε λοιπόν ε, συντονισμένη δράση για να προωθήσουμε τις επενδύσεις. Χρειάζονται περισσότερες, πιο βιώσιμες επενδύσεις και αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής αυτής. Οι επενδύσεις οδηγούν, αν δεν υπάρχουν μάλλον επενδύσεις, έχουμε λιγότερη ανάπτυξη, μειώνεται η ανταγωνιστικότητα κλπ. κλπ. Οι επενδύσεις λοιπόν χρειάζονται. Σήμερα έχουμε 15% χαμηλότερα από ό,τι θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση για να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Όπως είπα όταν παρουσίασα το παιδιτικό μας πρόγραμμα στις 26 Νοεμβρίου, σας είπα ότι δημιουργείται ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατηγική Σημασία Επενδύσεων. Στόχος του είναι να χρησιμοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικέ επενδύσεις και να μπορέσει να τους δώσει όθηση κάτι το οποίο δεν θα είχε γίνει χωρίς να υπάρχει το ταμείο αυτό. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν περισσότερη όθηση στις χώρες μέλη οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Το ταμείο αυτό θα λειτουργήσει ώστε να χρησιμοποιηθούν τα οικονομικά μέσα τα οποία είναι πιο κατάλληλα για την ενεργειακή διασύνδεση, για παράδειγμα, για την εκπαίδευση, για τις υποδομές και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως αντιλαμβάνεστε, Πρόεδρε και κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, εγώ δεν μπορώ να δεσμευτώ οικονομικά για συγκεκριμένα προγράμματα. Όλα τα προγράμματα πρέπει να ελεγχθούν ανάλογα με την οικονομική τους βιωσιμότητα. Η Task Force την προηγούμενη εβδομάδα εξέτασε 2.000 προγράμματα. Εννοείται ότι δεν είναι όλα νέα στρατηγική σημασία και οικονομικά βιώσιμα. Όμως Υπήρξαν πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα. Υποδομές, ενεργειακή διασύνδεση Φιλανδίας με τις Βαλτικές χώρες, εκπαίδευση στην Ιταλία, ε, νοσοκομεία στο Βέλγιο, για να σας αναφέρω μερικά μόνο παραδείγματα. Για να δημιουργηθεί το ταμείο αυτό χρειάζεται μία νομική πράξη, η οποία πρέπει με συναπόφαση να υιοθετηθεί. Η Επιτροπή λοιπόν τον Ιανουάριο του 2015 θα κάνει την σχετική πρόταση και προσβλέπουμε στη δικιά σας στήριξη ώστε να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί την Άνοιξη το ταμείο αυτό. Να εγκριθεί την Άνοιξη και να αρχίσει να λειτουργεί στα μέσα της επόμενης χρονιάς. Βασιζόμαστε επίσης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία θα αρχίσει να χρησιμοποιεί το τα χρήματα ήδη από την αρχή της επόμενης χρονιάς και έχει συμφωνήσει η ΕΤΕ με την βασική αυτή ιδέα. Έχουν υποθεί πολλά για το πώς τα κράτη-μέλη θα συνεισφέρουν στο ταμείο αυτό. Το νέο αυτό ταμείο είναι αυτόνομο, αλλά θα επηρέασει πολύ περισσότερο τα πράγματα εφόσον τα κράτη-μέλη συνεισφέρουν. Κάποιες χώρες-μέλη έχουν πει ότι έχουν αυτή την πρόθεση. Περιμένουμε λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις από αυτά και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο να εκδηλώσει την πρόθεσή του να συνεισφέρει. Όχι μόνο με λόγια, όχι μόνο παρόλε παρόλε, όχι, χρειαζόμαστε χρήματα. Από τη δικιά μου την πλευρά έχω πει ποια είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι υπέρ δηλαδή της συνεισφοράς αυτής κεφαλαίων από τις χώρες μέλη και βάσει των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τον Ιανουάριο θα υπάρξουν οι κατευθυντήριες γραμμές. Θέλω επίσης να σας διασφαλίσω ότι για να προχωρήσουν τα προγράμματα και να κριθούν βάσει της πραγματικής τους αξίας θα υπάρξει μια ανάλυση από εμπειρογνώμονες ανεξάρτητους όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα του κάθε προγράμματος που προτείνεται. Δεν θα υπάρξουν γεωγραφικά ή τομεακά κριτήρια ποσοστώσεις θα υπάρξει και τεχνική αρρωγή ώστε τα προγράμματα να προχωρήσουν και να μπορέσουν όλες οι χώρες να υποβάλουν τα προγράμματά τους. Και θα υπάρχει διαφάνεια ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορέσουν να δώσουν συνέχεια με αποτελεσματικότητα στα προγράμματά τους. Οι προσπάθειες αυτές θα συνοδευτούν από συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί το επενδυτικό πλαίσιο και να μην υπάρχουν πια εμπόδια στην ενιαία αγορά. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Θυμόσαστε το τρίγωνο το οποίο σας είχα περιγράψει όταν σας παρουσίασα το επενδυτικό μας πρόγραμμα. Δηλαδή δημοσιονομική υπαγίωση, μεταρρυθμίσεις και προϋπολογισμός. Αυτά τα τρία στοιχεία του προγράμματος δεν έρχονται σε αντίθεση το ένα με το άλλο. Αντίθετα, συνδυάζονται μεταξύ τους. Ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί στη συλλογική προσπάθεια που κάναμε να μειώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα. Όμως, το επίπεδο του δημοσίου χρέους σε ορισμένες χώρες μέλη εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό και ένα υψηλό χρέος εμποδίζει την ε, θέληση που μπορεί να έχουν ε, οι ιδιωτικοί επενδυτές να επενδύσουν στην Ευρώπη. Αναμένω λοιπόν και προσδοκώ αύριο το Συμβούλιο να στηρίξει απολύτως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει στην εφαρμογή όλων των στοιχείων που συνθέτουν το επενδυτικό πλαίσιο. Προσδοκώ επίσης το Συμβούλιο να μας στηρίξει με τη χρήση όλων των οικονομικών μέσων κατά την επόμενη ε, χρηματοδοτική περίοδο. Αυτό σημαίνει πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική χρήση των πόρων. Προσβλέπω επίσης και στην συνεχή στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, το άλλο σημείο που θα συζητηθεί αύριο στο Συμβούλιο είναι η Ουκρανία. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ε, εκλέχθηκε βάσει των προτινόμενων μεταρρυθμίσεων. Όντω, υπάρχει πρόγραμμα δράση τη κυβέρνηση και χαιρόμαστε για την αποφασιστικότητα τη κυβέρνηση εκεί να προχωρήσει σε πολιτικέ και οικονομικέ μεταρρυθμίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε μέλη πρέπει να συνεχίσουν να διευκολύνουν και να στηρίζουν το έργο τη κυβέρνηση εκεί. Οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν είναι τεράστιε. Πρώτα απ' όλα, η ειρήνη στον Τόνερτ και γενικότερα στο Ανατολικό Τμήμα έχουμε δει τον τελευταίο καιρό λιγότερη βία. Πρέπει να πετύχει πλήρως η εκεχηρία και να υπάρξει μια ειρηνευτική διαδικασία η οποία να ολοκληρωθεί. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην Ανατολική Ουκρανία και θα επιμείνουμε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία του Μίνσκ. Επίσης η Ουκρανία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση. Αυτό οφείλεται σε μακροοικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα. Σε αυτά τα δύσκολα πλαίσια λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει χωρίς προηγούμενο οικονομική στήριξη προκειμένου να ε, εφαρμοστούν τα διάφορα μακροοικονομικά προγράμματα. 760 εκατομμύρια σε δάνεια επίσης εκταμιεύτηκαν τους τελευταίους δύο μήνες μετά από τα 600 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν το καλοκαίρι. 250 εκατομμύρια επιπλέον μπορούν να εκμεταμιευθούν στις αρχές του 2015 εάν βέβαια υπάρχουν κατάλληλες πολιτικές ε, συνθήκες. Η Ουκρανία βέβαια θα χρειαστεί περισσότερη βοήθεια. Η αξιολόγηση του οικονομικού κενού της Ουκρανίας έγινε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Χρειάζεται 15 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον η Ουκρανία για να μπορέσει να προχωρήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει μόνο στα πλαίσια του δικού της προπολογισμού, βάσει της γραμμής του προπολογισμού που διαθέτει, η οποία έτσι κι έχει περιοριστεί, με ένα μικρό ποσό και πολύ μικρά περιθώρια ελιγμών για τους επόμενους, για, τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο, γιατί αν δώσουμε περισσότερα χρήματα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε άλλες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν τους επόμενους μήνες. Συνεπώς, πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες για 2, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Αν δεν μπορέσουμε εμείς, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν και να μας βοηθήσουν με κάποια ευελιξία στον προπολογισμό. Έπειτα, η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει την ενεργειακή προμήθεια της χώρας. Η Ουκρανία έχει ήδη παραγγείλει ένα δισεκατομμύριο <clears throat> κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να ελέγχει την εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσει να θαρρύνει την κυβέρνηση της Ουκρανίας για να μπορέσει αποτελεσματικά να προμηθεύεται από την Ρωσία φυσικό αέριο. Αυτά ήταν τα κυρία σημεία λοιπόν που ήθελα να σας αναφέρω πρόεδρε. Και θα δούμε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μετά τι στάση ευθύνη θα δείξουν και οι χώρες μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γιούγκερ από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ο πρόεδρο ε, τη ομάδα, ο κύριο Βίμπα. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε, mm. του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε λίγο πριν τι ε, εορτέ των Χριστουγέννων, ε, τι καλύτερε ευχέ μου λοιπόν. Και η πρώτη ευχή μου είναι προ το Συμβούλιο. μήπως θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτήν την μόνιμη συζήτηση για, το, για την ευελιξία και τη λιτότητα. Χρόνια τώρα τα συζητάει το Συμβούλιο. Ο Ζαν claude Juncker έχει κάνει καλές προτάσεις για να ξεπεράσουμε αυτή τη συζήτηση. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο επενδύσεων. Πρόεδρος, κύριε Βίμπε, υπάρχουν ε, προβλήματα με κάποιες γλώσσες. Α, με τα Ιταλικά, με τα Ιταλικά μάλιστα. η διερμηνία προς τα Ιταλικά είναι τώρα εντάξει. Εντάξει, εντάξει, ωραία, μπορείτε να συνεχίσετε. Το πρώτο, όπως είπα, είναι το πακέτο επενδύσεων. Ο Ζαν Κλοντ προτείνει μία νέα μέθοδο, τη συζητήσαμε αναλυτικά, όχι νέα χρέη, να αξιοποιήσουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο. 300 δις. Υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση. Με αυτό η Ευρώπη θα κάνει αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαίοι. Οπότε το θέμα είναι ενώπιον του Συμβουλίου τώρα. Και παρακαλούμε να υπάρξει στήριξη. Καλούμε για υποστήριξη. Χρειαζόμαστε αυτό το σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη. Και το εθνικό επίπεδο καλείται να συμβάλλει. Θα ήταν σκόπιμο όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη τις επόμενες μέρες να καταστήσουν ε, σαφές ότι θα συμβάλλουν. Και προς τη χώρα μου απευθυνόμενος θα ήταν καλό να συμβάλλει και η Γερμανία να στηρίξει το πακέτο το σύμφωνο επενδύσεων. Θέλουμε να δημιουργηθεί μια δυναμική και για τα 2.000 προγράμματα θέλω να πω ότι σκόπιμο θα είναι να συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί πολλά από τα προγράμματα αυτά είναι σαν ένας ε, κατάλογος επιθυμιών και όχι προτεραιότητες. Και προτεραιότητες χρειαζόμαστε για το μέλλον της Ευρώπης. Δεύτερον, δεύτερον αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πρόσκληση προς αυτούς που θέλουν ευελιξία και περισσότερο χρόνο να αξιοποιήσουν μέχρι το Μάρτιο, να δώσουν χρόνο μέχρι το Μάρτιο, χρόνο στην ε, πρόταση ε, Juncker. Δεν είναι απλώς μια προσφορά, είναι μια υποχρέωση να γίνουν οι αναγκαίες διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Να αξιοποιήσουν λοιπόν αυτή την ε, προσφορά Juncker. Θέλω να πω ότι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ένωσης, η Γαλλία, μας ε, δημιουργεί ανησυχίες γιατί στη Γαλλία συζητούν να είναι δυνατόν να ανοίγουν τα καταστήματα δύο Κυριακές ε, το μήνα συγγνώμη, το χρόνο για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν περισσότερο οι τουρίστες. Χρειάζεται πολύ σημαντικότερα θέματα να συζητηθούν, ούτω ώστε η δεύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης για να μπορέσει να ε, προετοιμαστεί καλύτερα για την παγκοσμιοποίηση. Μας ανησυχεί αυτό. Και πρέπει να τονίσω ότι χωρίς μια ισχυρή Γαλλία δεν έχει μέλλον η Ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, να πω κάτι ακόμη σε σχέση με αυτό. Τις τελευταίες μέρες έγιναν συζητήσεις για την Τρόικα στην Ελλάδα. Αν δούμε ε, τι απαιτούν οι Ευρωπαίοι εταίροι από την Ελλάδα που έκαναν τόσες προσπάθειες. Με τη στήριξη του Ιταλού και του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών πρέπει να ζητήσουμε αυτό που ζητάμε ε, στην Γαλλία και από την Ελλάδα. Και πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε δίκαιοι έναντι όλων των κρατών μελών. Πρέπει να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Γι' αυτό παρακαλώ ο καθένας να αξιοποιήσει την προσφορά που μας κάνει η Κομισιόν. Θα ήταν καλό εάν ε, η Γερμανία συμβάλλει στον Κορβανά και αν η Γαλλία κάνει τις αναγκαίες αλλαγές. Η ομάδα μας θα συζητήσει και θα έχει ως κέντρο της προσοχής της τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την Ευρώπη. Και γι' αυτό και με ευκαιρία την, συζήτηση για το πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν θέλω να τονίσω ότι υποστηρίζουμε τις προτάσεις ε, Τίμερμανς ο, έχει ο σοσιαλδημοκράτης κύριος Τίμερμανς την πλήρη υποστήριξή μας και για τα θέματα της φορολόγησης για τα οποία είχε τόσες αμφιβολίες η ομάδα των σοσιαλιστών. Νομίζω ότι οι προτάσεις που έχουν γίνει είναι πολύ καλές. Έχουν γίνει από έναν ε, σοσιαλιστή επίτροπο, τον κύριο Μοσκοβισή, και ελπίζω οι σοσιαλιστές να έχουν τόση εμπιστοσύνη στον Μοσκοβισή όπως έχουμε και εμείς. Πρέπει να το πω αυτό. Να τονίσω δύο άλλα σημεία. Το πρώτο είναι το TTIP, η Συμφωνία για Επενδύσεις και το Εμπόριο. Είναι πολύ καλό που το Συμβούλιο δήλωσε ότι μετά τις ε, συζητήσεις με την Αυστραλία που έγιναν στην Αυστραλία για το θέμα αυτό θα προχωρήσουμε τώρα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε δέσμευση. Θέλουμε βεβαίως να έχουμε υψηλές προδιαγραφές ως Ευρωπαίοι αλλά θέλουμε να προχωρήσει το παγκόσμιο εμπόριο. Γι' αυτό χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Συμβούλιο να προωθήσει το θέμα αυτό. Και τελευταίο, ένα θέμα που οπωσδήποτε μας ανησυχεί στην επικαιρότητα είναι εξελίξει εξελίξεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Τα είπε τα αναγκαία ο πρόεδρος Επιτροπής. Να πω μια φράση για τη Ρωσία. Αυτή τη βδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέβασε τα επιτόκια στο 17%. Το βασικό επιτόκιο. Το... Ε, αυτή η αύξηση σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να γίνουν πλέον επενδύσεις στο εσωτερικό. Το ρούβλι βεβαίως με αυτό σταθεροποιήθηκε για ένα διάστημα αλλά εξακολουθεί να πέφτει. Ε, βεβαίως ε, χαιρόμεθα που οι κυρώσεις έχουν αποτέλεσμα. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι ε, η πολιτική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η Μόσχα είναι λάθος για την ίδια της τη χώρα. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η προσφορά των Ευρωπαίων υπάρχει πάντα. Θέλουμε να έχουμε εταιρική σχέση με την Ρωσία και ελπίζουμε η Ρωσία να επανέλθει στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου που θα καταστούσε περιτές τις κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν ζητήσει πολύ μπλε κάρτα να πάμε με τη σειρά όμω. Η κυρία Μπερέσε, αν συμφωνεί ο κύριος Βέμπερ, θέλει να του κάνει μια ερώτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Βέμπερ, λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση και είμαι και εγώ υπέρ αυτής της μεταχείρισης. Όμως, για τις απαιτήσει μεταρρύθμισης προς τις χώρες που γνωρίζετε πολύ καλά, τι θα γίνει όπως η εργασία την Κυριακή, η εργασία των γυναικών, η καταπολέμηση της ένδυας. Τι απαντάτε στον κύριο Ντράγκη όταν μας καλεί να μιλήσουμε για τα συγκεντρωμένα αιτήματα των κρατών μελών και για τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα που θα μπορούσαν να καλύψουν κάποια κενά και που τόσο πολύ δεν αξιοποιούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνάδελφε Βερές, πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα για τι κυβερνήσει του ΕΛΚ στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Έχουν εισαγάγει διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Ο κύριο Ντομπρόφσκι στη Λετωνία, για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, στην Πορτογαλία, που σήμαιναν θυσίε, ε, σκληρέ θυσίε για τον πληθυσμό. Αν δείτε όμω τώρα την ανάπτυξη στην Ευρώπη, θα διαπιστώσετε ότι οι χώρες που προχώρησαν ε, σε μεταρρυθμίσεις, εφήρμοσαν μεταρρυθμίσεις, είναι η ατμομηχανή της ανάδειξης στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν έχει σπουδαία έννοια η ερώτησή σας. Αυτοί που θέλουν να καταπολεμήσουν την φτώχεια είναι αυτοί που έχουν το θάρρος να κάνουν τις διαστοτικές μεταρρυθμίσεις που οδηγούν τις χώρες τους στο μέλλον. Και σε αυτή την πολιτική θα μείνουμε. Για την ομάδα των Σελδημοκρατών ο πρόεδρος κ. Πιτέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, έχουμε μία επέτειο να γιορτάσουμε. Πριν από τέσσερα χρόνια, το 2010, ένας νέος από το τωρινό, Μάμετ Μπουασίση, ε, αυτοκτόνησε. Αυτοπυρπολήθηκε και από αυτό το γεγονός ξεκίνησε, ε, από αυτόν την ίσιο ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη. Ήταν 26 ετών και ήταν ένα άνεργο ο άνθρωπο αυτό. Πρέπει να πούμε ότι χωρί δουλειά κανεί δεν χάνει μόνο το εισόδημά του, χάνει την αξιοπρέπειά του, χάνει τον λόγο ύπαρξή του. Διότι η εργασία έχει μια ε, αξία αυτούσια που δίνει νόημα στη ζωή μα. Κάθε μέρα στην Ευρώπη 100 άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Πρόκειται για ένα πραγματικό δελτίο πολέμου. Η, μια ολόκληρη γενιά θυσιάζεται δεν μπορεί κανείς να υποκριθεί ότι δεν το βλέπει αυτό, ούτε θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα με ρητορικά τεχνάσματα. Θα πρέπει να δούμε την απογοήτευση και τον θυμό όσων δεν έχουν πια τίποτα να χάσουν, διότι ήδη έχουν χάσει την εξωπρέπειά τους. Αυτή η Ευρώπη υποφέρει και το λέω στον ε, κύριο Ντελαβέντοβα αυτό. Σε αυτήν την Ευρώπη λοιπόν που υποφέρει, σε αυτήν θα πρέπει να απευθυνθεί το Συμβούλιο αύριο. Θα πρέπει βεβαίω να πούμε ότι η παρέμβασή του πάει στη σωστή κατεύθυνση. Διότι οι επενδύσει όντω χρειάζεται να πάνε προ αυτό το στόχο και εκτιμούμε τους στόχους του προγράμματός σας, την αντιστροφή των τάσεων που υπήρχαν ως τώρα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Μάνφρεντ. Αυτή είναι η πραγματική προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο τους αριθμούς και τους λογαριασμούς. Ας σκεφτούμε τα άτομα, τους ανθρώπους που υποφέρουν. Για να μην υποφέρουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται επενδύσεις. Ανάπτυξη, βιωσιμότητα και δουλειές. Πρέπει όμως να φανούμε και συνεπείς ως προς το πρόγραμμα αυτό και μάλιστα να είμαστε και ταχείς να έχουμε σαφείς στόχους το ταμείο μας πρέπει να επικεντρωθεί στους, στις πιο ρηψοκίνδυνες επενδύσεις και στους πιο ενδιαφέροντες τομείς. Το είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ. Η καλύτερη, την καλύτερη απάντηση που μπορούμε να βρούμε στη Λίμα ή ε, την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Μέχρι τώρα είναι πολύ δειλά τα βήματά μας. Πρέπει να φανούμε αποφασιστικοί, με πυγμή και να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα λοιπόν πιο σταθερό με περισσότερους πόρους. Αυτό χρειάζεται να στηρίξουν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν φρέσκο χρήμα στο ταμείο αυτό. Καλά έκανε ο συνάδελφος Βέμπερ που ε, απίφθινε έκκληση και στη δική του τη χώρα. Όμως θα πρέπει να είναι ε, παρόμοιε οι συνεισφορέ των κρατών μελών προ το Ταμείο. Ιδάλω, κανεί δεν θα θέλει να το στηρίξει. Επίσης πρέπει να ξαναρχίσει η συζήτηση για την κοινή ανάληψη ευθύνης για τις συγχρηματοδοτήσεις των κρατών μελών προς τα προγράμματα που θα χρηματοδοτούνται από το ταμείο αυτό. Επίσης και η ευελιξία που χρειάζεται είναι ε, απαραίτητο στοιχείο για να δούμε το θέμα των κινήτρων που θα δώσουμε στα κράτη-μέλη. Κίνητρα για να στηρίξουν ακριβώς τα επενδυτικά προγράμματα του Ταμείου. Για να ε, λάβουν όλα αυτά σαρκα η Επιτροπή χρειάζεται τη στήριξή μας. Χρειάζεται τη στήριξη του Κοινοβουλίου μας. Στο Κοινοβούλιο αυτό δεν θα σας, ε, δε, στα πέντε περίσταση δεν θα σας αφήσουμε μόνους. Ούτε θα σας αφήσουμε να αποδυναμωθείτε όπως κάποιοι θέλουν ε, εκτός αυτής της ολομέλειας αλλά και ενδεχομένως εντός. Όμως ούτε κι εσείς πρέπει να μας αφήσετε μόνους. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στην επεξεργασία και την έγκριση του νέου Ευρωπαϊκού Στατηγικού Ταμείου και θα πρέπει να μπορέσει να εκφραστεί και για το πώς θα διαχειριστούμε το Ταμείο αυτό, ποια θα είναι η διακυβέρνησή του. Το Κοινοβούλιο λοιπόν βρίσκεται απέναντι ε, σε μια Ευρώπη που υποφέρει, αλλά εδώ πρέπει να πω ότι είναι απαράδεκτο το όπως έχουν τα πράγματα σήμερα το πρόγραμμα εργασίας να συζητια... στο πρόγραμμα εργασίας να συζητιάται μόνο η δημοσιονομική σταθεροποίηση και όχι το που θα βρεθούν κονδύλια για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ενώ δισεκατομμύρια διαφεύγουν από τα ταμεία των κρατών μελών με τη φοροδιαγωγή. Ε, η Ευρώπη για τους ισχυρούς είναι μια Ευρώπη που δεν την θέλουμε το πρόβλημα είναι οι επιχειρήσει που δεν πληρώνουν του φόρου. Δεν είναι απαραίτητα τα προβλήματα εκτό των συνόρων μα. Είναι αυτοί που περνάνε σε ενέργειε φοροαπάτη και φοροδιαφυγή. Αυτά τα θέματα πρέπει να απασχολήσουν το Συμβούλιο, κύριε Ντελαβέντοβα. Τα ε, συμπεριέλαβε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα εργασιών τη. Τα μέτρα που ζήτησα. Και ευχαριστούμε τον κύριο Τίμερμαν που τα ε, είδε αυτά τα θέματα, καθώ και τον κύριο Μοσκοβισή. Επίσης καταγράφω ε, τα σχόλια του κυρίου Βέμπερ για τον κύριο Μοσκοβισή, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ ούτως ή άλλως πάντοτε θα ε, ε, είμαστε αντικειμενικοί με οποιονδήποτε επίτροπε κάνει σωστά τη δουλειά του ε, ή οποιοδήποτε αντιπρόεδρο της, της Επιτροπής. Όπως είπε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, αυτή είναι μια νέα αρχή. Ολοκληρώνω, Πρόεδρε. Είναι μια νέα αρχή, αλλά για να είναι πραγματικά μια νέα αρχή πρέπει να δουλέψουμε εντατικά, με πάθος και πυγμή. Ευχαριστώ. <clears throat> Κύριε Πιτέλα, υπάρχει μια ερώτηση από πλευρά τη συναδέλφου Τζούλια Μούλ προ εσά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ρωτήσω τον κύριο Πιτέλα που είπε στην ομιλία του ότι ζητάμε χρήματα. Φυσικά, όχι κρατικά κονδύλια, ούτε των πολιτικών φίλων σας. Εσείς Πώ μπορείτε να ζητάτε περισσότερα χρήματα από του Ιταλού ή του Ευρωπαίου που αυτή τη στιγμή έχουν τσακιστεί στη δουλειά για να μπορούν να σα συντηρούν και να σα πληρώνουν στην Ιταλία. Προέκυψε σκάνδαλο όπου φάνηκε ότι για χρόνια το κόμμα σα αλλά και η δεξιά και η αριστερά ταυτόχρονα έκλεψαν εκατομμύρια ε, από του φτωχού μετανάστε. Στη Μόζε στη Βενετία, στην Έξπο του Μιλάνο. Αυτά που καλύφθηκαν χθε το βράδυ και τώρα ζητάτε κρατικά κονδύλια θα πρέπει να ντρέπεστε. Συνάδελφε, νομίζω ότι είναι ένα σχόλιο για σας την ίδια το πνεύμα της παρέμβασής σας. Δεν θα πω πολλά λόγια. Απλώς όταν ε, χρησιμοποιεί κανείς τέτοια στοιχεία ουσιαστικά παραπληροφορεί τους πολίτες. Ε, το ποιος έκλεψε ε, ανελαίητα για όλους θα φανεί. Οι κλέφτε βρίσκονται παντού και θα πρέπει να του καταπολεμήσουμε από κοινού. Είμαστε ένα κόμμα και μια μεγάλη πολιτική οικογένεια που αγωνιζόμαστε κατά τη διαφθορά, τη επεξαίρεση χρημάτων, κατά τη μαφία, κατά των εγκληματικών ομάδων, των ομάδων οργανωμένου εγκλήματο και των κακών πολιτικών. Όταν ζητούμε περισσότερα χρήματα, τα ζητάμε για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Ευχαριστώ πολύ. κύριε ο Και τώρα για την ομάδα ECR ο πρόεδρος Καμάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών χαιρόμεθα που κάποιος κάνει τα σωστά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Πώς θα υπάρξουν επενδύσεις. Δεύτερον, πώς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε αυτούς που είναι υπέρ της ε, αυτοδιάθεσης της ε, χώρας του στην Ουκρανία οι συναδελφοί μου θα μιλήσουν γι' αυτό. Χαιρετίζουμε τι προτάσει για το πρόγραμμα επενδύσεων, όχι για το περιεχόμενο, αλλά θα βοηθήσει να ξεκινήσει τη συζήτηση. Όχι απλώ μια συζήτηση για τα 315 δι, αλλά μια συζήτηση γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια ιδιωτικών επενδύσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλά δεν χρησιμοποιούνται ιδιωτικών επενδυτών. Πρέπει όμω ε, να τεθούν ερωτήματα. Ποιε θα είναι οι προτεραιότητε του επενδυτικού ταμείου, όπω ρώτησε ο Μάνφρεντ πώς θα μοχλεύσει τις ιδιωτικέ επενδύσεις. Πώς το Ταμείο αυτό θα αποφύγει καταστάσεις όπου ε, εθνικοποιούμε τις ζημίες και ιδιωτικοποιούμε τα κέρδη. Αλλά η συζήτηση που γίνεται τώρα για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις πρέπει να μετατραπεί σε πράξεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια αγορά για κεφάλαια, αγαθά και υπηρεσίες. Αλλά δεν τα έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ξεκινήσει την ενιαία αγορά για τα κεφάλαια. Αλλά δεν θέλουμε αυτή η ενιαία αγορά κεφαλαίων να είναι απλώς όλο και περισσότερες ρυθμίσεις. Θέλουμε να είναι ανοιχτή και διαφανής, να λειτουργεί σωστά, ούτω ώστε οι επιχειρήσεις να μην χρειάζεται να περιμένουν τόσο πολλά από τις τράπεζες. Πρέπει να σταματήσουν τα εμπόδια για τις επενδύσεις, όχι μόνο για ιδιωτικές επενδύσεις γενικά, αλλά ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομέ, σε μικρομεσαίε επιχειρήσει, ούτω ώστε οι καινοτόμε ιδέε να γίνουν πραγματικότητα. Γιατί η μη τραπεζική χρηματοδότηση, όπω τα κεφάλαια υψηλού κινδύνου, δεν χρησιμοποιούνται αρκετά στην Ευρώπη. Να σα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Συμμετέχω σε, ε, πολύ συχνά ε, σε ένα site που λέγεται Kiver, το οποίο βοηθάει επιχειρηματίες να ε, ξεκινήσουν επενδύσεις. Εγώ δανείζω σε αυτό το κεφάλαιο 25 ε, ευρώ κάθε τόσο, αλλά γιατί εγώ μπορώ να δανείσω 25 δολάρια ή 25 λίρες σε έναν επιχειρηματία σε μια φτωχή χώρα και δεν μπορώ να το κάνω στην ίδια μου τη χώρα. Πρέπει να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Προσπαθώντας να καταλάβω γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, κατάλαβα ότι δεν χρειαζόμαστε κρατικές παρεμβάσεις. Κατάλαβα ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο παρά να δώσουμε τη δυνατότητα να συλλέγονται χρήματα από το κοινό, ότι υπάρχουν χρήματα και απλώς πρέπει να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες να αξιοποιήσουν οι δανειστές τις τα μικρά ποσά που θέλουν να δανείσουν για να βοηθήσουν επενδυτικά προγράμματα έστω και μικρά. Όλα αυτά όμως δεν πρέπει να γίνουν μονομένα, πρέπει να είναι στα πλαίσια ενός παγκόσμιου πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Το Συμβούλιο επανέλαβε τις δεσμεύσεις του ότι θα αντιμετωπίσει τι ενεργειακέ προκλήσει για την Ευρώπη, ότι θα αναπτύξει την ψηφιακή ενιαία αγορά και ότι θα καταλήξουν οι διμερεί εμπορικέ διαπραγματεύσει. Για όλα αυτά τα θέματα η ομάδα μου έχει ξεκινήσει ομάδε εργασία για να παρουσιάσουν νέε ιδέε. Συμφωνούμε, αλλά όχι μόνο συμφωνούμε, θα σα βοηθήσουμε με τι δικέ μα ιδέε να αντιμετωπίσετε αυτέ τι προκλήσει. Αλλά δεν έχει καμία έννοια οι Ευρωπαίοι ηγέτε στι Βρυξέλλε να λένε ότι πρέπει να υπάρχει νοοτροπία ανταγωνισμού για να βοηθήσουμε τι ιδιωτικέ επενδύσει και μετά να επιστρέφουν στι πρωτεύουσέ του και να μην, να μην παίρνουν τι δύσκολε αποφάσει που πρέπει να πάρουν. Πολλέ από αυτέ τι ε, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει πρέπει να τι κάνουμε παρά το ότι δεν είναι δημοφιλεί. Και ξέρουμε ότι τα υπάρχοντα συμφέροντα θα, θα τι ε, προσπαθήσουν να τι ε, σταματήσουν. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε. Εγώ θέλω να πάρω κάποιε αποφάσει για τον νέο χρόνο. Η πρώτη μου θα είναι να κάνουν περισσότερη γυμναστική και οι ηγέτες του Συμβουλίου να πάρουν τη δική τους απόφαση, να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες τους, να σταματήσουν τα εμπόδια στις επενδύσεις, να σταματήσουν να μειώσουν τη γραφειοκρατία, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Και ας ελπίσουμε ότι το 2015 να είναι η χρονιά όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξαναρχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Καλή χρονιά σε όλους. Κύριε Καμάλ, ο κύριος Κόμπερν θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Το δέχεστε? Παρακαλώ. Ο κύριος Κόμπερν. Κύριε Καμάλ, συμφωνείτε ότι τα ισχυρότερα κράτη της Ευρώπης είναι αυτά που είναι εκτός του ευρώ και που καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το επιχειρηματικό πνεύμα. Κάτι τέτοιο μπορεί να μην το καταλαβαίνετε εδώ μέσα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπαθεί να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και όχι να κάνει κρατικές επενδύσεις. Οι κυβερνήσεις δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας. Και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το καταλαβαίνει αυτό, μήπως θα ήμασταν καλύτερα κύριε Καμάλ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμάλ, κύριε Κόμπερν, κύριε Κόμπερν, κύριε Κόμπερν, Πρώτα απ' όλα, αναρωτιόμουν πότε θα μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Και δεύτερον, δεν με εκπλήσει η ερώτηση. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι εξεπλάγει κανεί από την ερώτηση που κάνατε. Κοιτάξτε κύριε Κόμπερν, η πρώτη σας ερώτηση ήταν γιατί οι χώρες εκτός Ευρωζώνης προκαλούν περισσότερες επενδύσεις. Ξέρω ότι διαβάζετε τις προηγούμενες ομιλίες μου και θα διαβάσατε σε μια προηγούμενη ομιλία ότι είπα ακριβώς αυτό. Οπότε το δίδαγμα για την Ευρωζώνη είναι να καταλάβει γιατί δεν μπορεί να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις. Ελπίζω να γίνει αυτό τα επόμενα χρόνια. Και τώρα για τους φιλελεύθερους ο πρόεδρος κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Την παρέμβασή μου δεν θέλω να την κάνω τόσο προς την Επιτροπή, αλλά προς το Συμβούλιο. Γιατί η Επιτροπή έχει παρουσιάσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια φιλόδοξη απάντηση, ανταπόκριση από το Συμβούλιο αύριο και μεθαύριο, και πέμπτη μάλλον και Παρασκευή. Κύριε Τελεβέντοβα, πρέπει να σας πω ότι εγώ είδα το σχέδιο συμπερασμάτων. Κόλλα light, ξέρετε τι είναι. Ε, εδώ θα έλεγα Council light. Τα συμπεράσματα δηλαδή του Συμβουλίου που θα βγουν τις επόμενες μέρες αυτό θυμίζουν. Εντάξει, όχι μηδέν, όχι zero κόλλα, όχι, εντάξει. Δεν λέω ότι θα είναι μηδενικά. Light όμω θα είναι. Και έχω την εντύπωση ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν αντιλαμβάνονται καν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Λένε καλούμε, στηρίζουμε, ξανακαλούμε, ξαναστηρίζουμε. Μια συνεχής πρόσκληση είναι για συμμετοχή. Όμως θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ε, αναλάβετε αποφάσεις σε σχέση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να προωθηθεί το φιλόδοξο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, πρέπει να αποφασίσετε με τις 28 χώρες μέλη να μπείτε σε αυτό το σχήμα εγγύσεων του επενδυτικού ταμείου. Αυτό. Όχι προσκαλούμε, κάνουμε, σκεφτόμαστε. Όχι, τώρα πρέπει να πάρετε την απόφαση 28 χώρες μέλη για τη συμμετοχή σας στο επενδυτικό αυτό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν χρειάζεται να αλλάξει το πρόγραμμα σταθερότητα. Μπορείτε κάλλιστα να το κάνετε με του σημερινού κανόνε. Δεύτερον, να ενισχύσετε το Ταμείο με εθνικέ συμμετοχέ μέσω ε, φορολόγηση του Ταμείου αυτού. Πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε έτσι να έχουν αυτή την ε, όθηση να επενδύσουν. Τρίτον, πρέπει να αποφασίσετε πιέσαστε να πείτε ότι η πρώτη επένδυση θα πάει σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα και την άλλη που όντως έχουν προχωρήσει σε θετικές μεταρρυθμίσεις. Είναι ένα θετικό κίνητρο για αυτές τις χώρες να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις. Έπειτα το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Πώ θα βγούμε από την κρίση, λέτε. Ε, μα αποφασίστε για το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Εδώ και μήνε το έχετε στο τραπέζι του Συμβουλίου. Και τι κάνετε, μόνο πίσω πάτε δεν ε, μας απαλλάσσετε από τα τέλη περιαγωγής, δεν προωθείτε την εναρμόνιση, τίποτα. Ε, να αποφασίσετε επιτέλους για το πακέτο αυτό, το οποίο πάνω από ένα χρόνο το έχετε στη δικιά σας την πλευρά. Έτσι θα ενισχυθεί η ψηφιακή αγορά της Ευρώπης. Πέμπτο, να αποφασίσετε ένα δεύτερο πακέτο για τα ψηφιακά. Το χρειαζόμαστε οι μισές ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Spotify ούτε το Netflix. Γιατί, Γιατί δεν υπάρχει ένας ρυθμιστής και ένα καθεστώς ε, copyright. Έπειτα, η ενεργειακή κοινότητα και αυτή πρέπει να προωθηθεί από εσά. Το Συμβούλιο εμποδίζει να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Και τέλος αυτό που είπε και ο κύριος Καμάλ. Επιτέλους αντελήφθηκε ο κύριος Καμάλ τα πλεονεκτήματα από μια ενωμένη Ευρώπη, γιατί αναφέρθηκε στις κεφαλαϊκές αγορές. Όντως, δεν έχουμε μια πιστοτική αγορά. Όχι, είναι κατακαιρματισμένη στην Ευρώπη. Αν έχετε ένα κεφάλαιο σε μια χώρα, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε μια άλλη χώρα. Αυτές λοιπόν είναι αποφάσεις που πρέπει να προωθήσετε και όχι αυτά τα ψευτοσυμπεράσματα που βλέπω εδώ, Μα αν λάβετε υπόψη σας πόσο βαθιά είναι αυτή η κρίση, πόσο πολύ μας λείπουν οι επενδύσεις από το 2008 και μετά, εγώ αυτό που περιμένω από το Συμβούλιο, όχι μόνο από την Ιταλική Προεδρία, αλλά από τις 28 χώρες μέλη, είναι επιτέλους για πρώτη φορά να πάρουν συγκεκριμένες ε, αποφάσεις για να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας βοηθήσουν στην Ευρώπη να βγούμε από την κρίση. Αυτό είναι που ζητάω. Ξέρω ότι εσείς πρόεδροι είστε εδώ. Ξέρω ότι πάντα από την αρχή ζητάτε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να περάσει αυτό το μήνυμα. Ελπίζω λοιπόν και αύριο στο Συμβούλιο να κάνετε το ίδιο κύριε Πρόεδρε, να πάτε στο Συμβούλιο και να περάσετε αυτό ακριβώ το μήνυμα ότι πρέπει να μας βγάλουν από αυτή την κρίση επιτέλους. Κύριε ε, Φερχόφστατ, υπάρχει μια ερώτηση του κύριου Στόιχατ προς εσάς. Παρακαλώ. Κύριε Φερχόφστατ, είστε τυπικά επικεφαλής των φιλελευθέρων, της φιλελεύθερης ομάδας. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί πάντα καλείται το κράτος, γιατί πάντα πρέπει για όλες αυτές τις επενδύσεις να αποφασίζει το κράτος, όχι επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα επενδύσεων 315 δις γιατί πρέπει να το αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη γιατί δεν θα πρέπει απλώς να δώσουν εγγυήσει στα κράτη γιατί από ό,τι φαίνεται για τους ε, ιδιωτικούς επενδυτές είναι πολύ υψηλό το κόστος πώς είναι δυνατόν εσείς ως φιλελεύθερος να καλείτε πάντα για παρέμβαση του κράτους Στις προτάσεις της Επιτροπής δεν αναφέρονται κρατικά κονδύλια ιδιωτικά αναφέρονται ε, δεν το έχετε καταλάβει το μόνο το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι χώρες μέλη είναι ότι εγγυώνται ένα πρώτο κομμάτι. Αν τυχόν κάποια από αυτές τις επενδύσεις πάει στραβά. Αυτό είναι που γίνεται και αυτό είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο. Όλοι οι θεσμικοί επενδυτές μας συμφωνούν ότι πρόκειται για συνεργασία ανάμεσα στην εγγύηση των χωρών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά ιδιωτικών επενδύσεων. Περί αυτού πρόκειται. Δεν πρόκειται για δημόσιο χρήμα. Είμαι φιλελεύθερος, είμαι υπέρ του ιδιωτικού χρήματος. Ευχαριστώ για την ενία αριστερά η πρόεδρος κυρία Τσίμα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να στραφώ και εγώ προς το Συμβούλιο. Για μένα τίθεται το ερώτημα το πρώτο λοιπόν θέμα τι έχει αλλάξει μετά τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών Ενόψεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι διαπιστώνουμε. Υπάρχει ετοιμότητα των εκπροσώπων των κρατών να υπάρξουν βιώσιμες επενδύσεις για να υπάρχουμε μια ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και να θέσουμε προτεραιότητες για τις επενδύσεις αυτές. Αυτό είναι το κύριο. Δεν το βλέπω αυτό. Και αυτό είναι ακριβώς η ουσία του προβλήματος. Ο κύριος Γιούνκερ ως πρόεδρος της Κομισιόν μας παρουσίασε ένα πρόγραμμα της Κομισιόν που κυρίως θα έπρεπε να βοηθήσει κοινωνική, βιώσιμη, οικολογική, οικονομική ανάπτυξη στα κράτη-μέλη. Έχω την εντύπωση όμως ότι όπως η κυρία Στόρχ δεν κατάλαβε τώρα το περιεχόμενο του επενδυτικού προγράμματος, έχει απόλυτο δίκιο, δεν το κατάλαβε. Για μένα το παράλογο είναι ότι παρά το ότι δεν το κατάλαβε το πρόβλημα, αντέστρεψε την κατάσταση. Και είπε βεβαίως ότι όλα πρέπει να είναι ιδιωτικές επενδύσεις ότι δεν πρέπει να γίνονται κρατικές επενδύσεις. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστιο πρόβλημα ότι δεν γίνονται οι αναγκαίες βιώσιμες επενδύσεις μέσω προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων. Και γι' αυτό είμαι πλήρω αντίθετη με τις θέσεις ε, του κόμματο ε, Εναλλακτική για τη Γερμανία. Γιατί λοιπόν λέτε ότι τόσο μικρή είναι η εμπιστοσύνη που έχετε προς τους ε, αρχηγούς των κρατών μελών που δεν πιστεύετε ότι μπορούν να κάνουν δημόσιες επενδύσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Γκάμπριελ είπε ότι για αυτόν όλα αυτά είναι μαύρη μαγεία, βουντού η λέξη που χρησιμοποίησε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά ακόμη αν θέλουμε να υπάρξει βιώσιμη κοινωνική πολιτική που να δημιουργήσει απασχόληση. Εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει κοντά σε αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει ήδη ένας κατάλογος και θα ήθελα να μάθω πώς ε, πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι υπάρχει ένας κατάλογος, ένας κατάλογος μείωσης των δικαιωμάτων. Πώς να βοηθήσουμε τις επενδύσεις όταν καταργούμε την άδεια τη γονική άδεια. Πώς ε, θα προωθήσουμε τις επενδύσεις όταν μειώνουμε τις οικολογικές προδιαγραφές, τις οποίες όλοι έχουμε συμφωνήσει δημοκρατικά. Όλα αυτά αφαιρούνται από τη συζήτηση. Για παράδειγμα έχουμε το πρόγραμμα για τον καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα, το οποίο δεν προωθούμε. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτές οι μειώσεις που κάνουμε θα έχει ελάχιστες επιπτώσεις αλλά θα έχει ως επίπτωση ότι μειώνονται οι οικολογικές και κοινωνικές προδιαγραφές στα κράτη-μέλη. Γιατί, για παράδειγμα, τα προγράμματα τα οποία συλλέξατε τώρα δεν έχουν ήδη προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις. Αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, πρέπει να αλλάξουμε τις προϋποθέσεις σε εθνικό επίπεδο. Επ' αυτού πρέπει να είμαστε σαφείς. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Τσίμα, η κυρία Φωνστόρ θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Βλέπω ότι η κυρία Στόρχ θέλει σήμερα να μας ε, αποδείξει πόσα γνωρίζει. Θέλετε να κάνετε ερώτηση κυρία Στόρχ. Δεν κατάλαβα αν είπατε ναι, νόμιζα ότι εκφράσατε αμφιβολίες. Αν σας κατάλαβα καλά, πώς θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει το πρόγραμμα επενδύσεων. Χρειάζονται 21 δις δημόσιες ε, πιστώσεις που θα είναι οι ε, εγγυήσεις για τους ιδιωτικούς επενδυτές. Φαίνεται λοιπόν δεν θέλουν να ε, επενδύσουν. Γιατί δεν ενδιαφέρονται, δεν θέλουν να κερδίσουν χρήματα. Πώς εξηγείτε ότι αυτά τα 21 δισεκατομμύρια δημοσίων πόρων Θέλουμε να τα κάνουμε τελικά 66 δισεκατομμύρια ε, πιστώσεων για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδυτέ. Πού είναι η λογική αυτή, κυρία Στόρχ, λέει η κυρία Τσίμερ. Το ερώτημα αυτό να το θέσω στον κύριο Γιούνκερ και όχι σε μένα. Ευχαριστώ για την ομάδα των Πρασίνων η πρόεδρος κυρία Χάρμς. Λοιπόν, να επανέλθω σε αυτά που υπόθηκαν. Ε, να επανέλθω συγκεκριμένα σε αυτά που είπε ο κύριος Φερχόφστατ στο σχέδιο ψηφίσματος διαπιστώνω ότι με την ανάληψη από τον κύριο Τούσκ του Συμβουλίου βλέπω ότι είναι, περιέχονται πολλές ε, προσπάθειες να ε, κάνουμε ευχολόγια. Δεν βλέπω καμία διάθεση του Συμβουλίου να αποκτήσουμε ένα μόνιμα σταθερό ευρώ, να ξεφύγουμε από την κρίση. Όλα τα μέτρα που προτείνονται δεν περιέχουν μια κοινή οικονομική πολιτική, την οποία χρειαζόμαστε για να σταθεροποιήσουμε το ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα αξιοποιήσετε όλα αυτά τα μέτρα. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο επικρατεί άποψη ότι έναντι των πολιτών ε, δεν τολμούν καν να ε, αναφέρουν τέτοιες ιδέες. Πώς λοιπόν θα δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης. Διαβάσατε τι έγινε με τις διαρροές για το Λουξεμβούργο, το LuxLeaks και τις επιπτώσεις του. Τι αποτέλεσμα είχαν ότι δεσμεύεται τώρα το Συμβούλιο ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώνουν φόρο εκεί που έχουν τα κέρδη. Αυτό είναι ένα μέτρο που αν το εφαρμόζατε θα μπορούσατε αμέσως από τη μία μέρα στην άλλη να επανακτήσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Έχω την εντύπωση όταν βλέπω αυτό το σύντομο σχέδιο αποφάσεων του Συμβουλίου βλέπω ότι οι πηγές χρηματοδότησης θα είναι διάφορες. Έχω την εντύπωση ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι μέσω ελευθέρου εμπορίου και την κατάργηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαρφών θα μπορέσουμε να προωθήσουμε μεγάλες επενδύσεις και έτσι να δημιουργήσουμε απασχόληση. Εγώ όμως δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω, κύριε Γιούνκερ και κύριε Τούμερμανς, ότι πρέπει να κάνετε τεράστιες προσπάθειες, διότι έχει, υπάρχει απλώς ένας κατάλογος είναι ένας κατάλογος ε, χριστουγεννιάτικων δώρων, ιδιαίτερα μακροσκελής. Κύριε Τίμερο, είστε γνωστός ως σκληρός διαπραγματευτής. Πρέπει να εγκρίνετε μόνο προγράμματα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος επενδύσεων που είναι πραγματικά κατάλληλα για βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη. Και σας παρακαλώ να φροντίσετε να μην ε, προωθήσουμε την ε, πυρηνική βιομηχανία η οποία μετά από 40 χρόνια ακόμη δεν ανταγωνιστική μέσω ε, τρομερών επιδοτήσεων να αναστηθεί και πάλι. Θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων είναι τόσο φορτωμένο από προγράμματα από το παρελθόν. Ήταν καλή ιδέα αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων. Ελπίζω όμως να εφαρμοστεί και σωστά. γιατί η Ρωσία τώρα καλύτερα στο κείμενο του Συμβουλίου να μην μιλάμε για την Ουκρανία μόνο, να πούμε ότι υπάρχει βαθιά κρίση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και, Τουρκία, και Ρωσίας. Αυτό το μαθαίνουμε από τις ειδήσει των τελευταίων ημερών. Δεν εξαρτώμεθα μόνο εμείς από τις εισαγωγές ενέργειας. Η Ρωσία είναι σε πολύ διαφορετική κατάσταση από την κατάσταση του ψυχρού πολέμου. Τώρα είναι πολύ στενά διασυνδεδεμένη με την Ευρώπη. Όλα όσα αποφασίσαμε μέχρι τώρα είναι σωστά για την ε, Ρωσία. Δεν θα πρέπει να διασπαστεί το Συμβούλιο οποιασδήποτε προσπάθειε και γίνονται από πλευρά τη Μόσχα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρο. Υπάρχει μία ερώτηση ε, ε, του βουλευτού Εύερης προ εσά. Τη παρακαλώ. Ο κύριος Average. Ο κύριος Καλημέρα σας και καλά Χριστούγεννα. Απλώς επειδή μιλήσατε για την ενεργειακή βιομηχανία και τις επιδοτήσεις, δηλαδή συμφωνείτε μαζί μου ότι με όλες αυτές τις πηγές παραγωγής ενέργειας που είναι τόσο αναποτελεσματικές και δεν υπάρχει αποδοτικότητα, θα πρέπει να επιδοτούμε με τις ε, γεννήτριε ενέργειας, ενέργεια, με τι ανεμογεννήτριες. Τι επενδύσεις πιστεύετε ότι χρειάζονται, μήπω μόνο ε, να επενδύσουμε εκεί που υπάρχει πραγματικά αποτέλεσμα. Ναι, κοιτάξτε στην Μεγάλη Βρετανία, εάν πιστεύετε ότι είναι ανταγωνιστική η πυρηνική βιομηχανία, τότε δεν θα έπρεπε να προτείνετε επιδοτήσει για αυτά τα προγράμματα. Και δεύτερον, δεν θα πρέπει να καθορίσετε εγγυημένη μόνιμη τιμή για το ρεύμα που παράγεται για παράδειγμα στο Hinkley Point είναι εγγυημένη αυτή η τιμή για 35 χρόνια και επίσης είναι και τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενη και ήδη σήμερα είναι πιο ακριβή από την ε, ε, εντός των ακτών ε, αιωλική ενέργεια. Αλλιώς θα επιτύχουμε ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα για το EFTD ο κύριος Νάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν δει κανεί την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου αυτού, μα θυμίζει τα ίδια παλιά θέματα τη ανάπτυξη και τη απασχόληση. Λε και τα θέματα αυτά ξανασυζητιούνται διαρκώ και δεν γίνεται τίποτε. Στην Ισπανία πάνω από 50% ενεργεία των νέων, η, Γαλλία της, ε, η οικονομία της Γαλλίας ε, συρρυκνώνεται και η Ελλάδα δεν μπορεί ακόμη να τονώσει την οικονομία της. Όμως, ασχέτως με το εάν πάρετε τις σωστές ή τις λανθασμένες αποφάσεις, δεν φαίνεται να λύνεται κανένα πρόβλημα. Ακόμα και με το πρόγραμμα Juncker φαίνεται σαν να έχουμε μαγικά από 21 εκατομμύρια ε, μία μετατροπή σε 315 μου θυμίζεται ένα παλιό λαϊκό τραγούδι, ένα παραμύθι στη Νέα Υόρκη, το αμερικανικό όνειρο. Αυτό φαίνεται να ζούμε σήμερα στο Στρασβούργο. Κύριε Juncker. Ξέρω ότι σας αρέσει και να πίνετε και να καπνίζετε. Αλλά ελπίζω ότι σας αρέσει και να είστε προσγειωμένος και να σας αρέσει να παραμένετε συνεπείς. Εδώ μιλήσαμε για θέσεις απασχόλησης. Όμως φαίνεται να υπάρχει ένας αγώνας εδώ, ένας εναγωνισμός σαν υποδρομία στην Ευρώπη και αυτό που ζούμε φαίνεται σαν όνειρο πλέον. Όμως υπάρχει ένας ωραιότερος αγώνας απόψε που θα μπορούσαμε να το, να, θα μπορούσατε να το σκεφτείτε λόγω του τίτλου. Το ονομάζεται μια ε, super fantasy, δηλαδή είναι μια φαντασίωση αυτό που ζούμε. Είναι οικονομικοί υπολογισμοί που ξεπερνούν τη φαντασία αυτή που κάνετε. Οι εκτιμήσεις σας ε, είναι ε, τελείως απάσιμες βάσει της σημερινής τη ω τώρα πείρα μα. Δεν σα πιστεύουμε πια, γιατί οι ίδιοι τεχνοκράτε τη Ευρώπη μα είπατε με το πρόγραμμά σα πριν 10 χρόνια ότι θα, δημιουργηθεί, ε, θα δημιουργηθούν δουλειέ και απασχόληση. Όμω καταραίουμε στην, στο διεθνή ανταγωνισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να είναι η απάντηση, κυρίε και κύριοι. Το επενδυτικό σα πρόγραμμα φαίνεται να είναι απλώς ένα, μια ε, ένα μεγάλο τέχνασμα και μια μεγάλη γαλοπούλα χριστουγεννιάτικη που μου δίνει την ευκαιρία να σας πω και καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Κύριε Νάτολ, ο συνάδελφος Γιάκον Σάρη θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Δέχεστε? Ε, η κυρία Γιάκον Σάρη, παρακαλώ. Κύριε Νάταλ, Μόλις μας είπατε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής και το επενδυτικό πρόγραμμα είναι αυτό που πάντα ήταν η ομιλία σας, όμως το ίδιο. Ε, και εσείς επαναληφθήκατε. Μιλήσατε για υποδρομίες και στοιχήματα αντί για επενδύσεις. Όμως Κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει στην ονομασία της ομάδας σας. Έχει προσθεθεί ένα γράμμα στο ακρόνιμο. Τι προτείνετε εσείς εναλλακτική, τι προτείνετε για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, για έχουμε πάλι απασχόληση. Κοιτάξτε, κάποιε φορέ στον υπόδρομο, όποιο στοιχηματίζει στα έστα κάποια άλογα, καμιά φορά κερδίζει κιόλα. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι ότι η εναλλακτική είναι μια ελεύθερη ε, Ευρώπη με ανεξάρτητα κάτι μέλη που λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Αυτό που δεν θέλουμε είναι ένας οργανισμός τελείως τεχνοκρατικός με αποφάσεις που να λαμβάνονται από μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πίσω από κλειστέ πόρτε λαμβάνει αποφάσει χωρί δημοψηφίσματα, χωρί καμία δημοκρατία. Εμεί θέλουμε τη δημοκρατία, την ελευθερία και γι' αυτό είμαστε η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Δεγκράφ ε, μη εγγεγραμμένος. Ο κύριος Γιούγκερ μας προτείνει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό σημαίνει ότι η Ολλανδία πρέπει να δώσει άλλα 8 δισεκατομμύρια να ταρπάξει ουσιαστικά από τους πολίτες της. Για να φτιαχτούν αεροδρόμια όπου δεν πατάει ψυχή, για να φτιαχτούν ε, προστατευτικά για τον ήχο σε δρόμους όπου δεν κατοικεί κανείς και για να πληρωθούν ανόητα ενεργειακά προγράμματα. Θα κλείσει συμφωνίες, θα παρασκήνει ο κύριος Γιούνκερ όπως έκανε και όταν ήταν πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Το αρχικό ποσό των 21 δισεκατομμυρίων πρέπει να, που θα δώσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΤΕ θα πρέπει να καταλήξουν σε 300 δισεκατομμύρια μέσω επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Έχει προβλέψει φορολογικές διευκολύνσεις ο κύριος Γιούνκερ για τις επιχειρήσεις. Ή πιστεύει ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την ψευδέστηση, το Φάτα μια, μιας μεγάλης ευρωπαϊκής αυτοκρατορίας, ενώ υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στην οικονομική κατάσταση των χωρών μελών. Το τίμημα της αυτοκρατορίας αυτό όμως το πληρώνουν οι πολίτες μέσω αματηρών οικονομιών, μέσω βαριάς φορολογίας, μείωση της ευημερία τους και χάνοντα τι θέσεις απασχόλησής του στη δουλειά του. Αντί για αυτό το ανόητο πρόγραμμα ο κύριος Γιούγκερ και το Συμβούλιο θα έπρεπε μάλλον να διαλύσουν την Ευρώπη και το ευρώ ώστε να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία, οι χώρες μέλη να μπορούν να αποφασίζουν για τη δικιά τους ευημερία, να έχουν το δικό του νόμισμα που να αντιστοιχεί στη δικιά του οικονομία και να κρατάμε και του μετανάστε ε, μακριά ε, μια που είτε μα κοστίζουν δισεκατομμύρια είτε κινδυνεύει η ασφάλειά μα από τζιχατιστέ. Αυτά θα έπρεπε να κάνουν, ο κ. Γιούνκερ, αλλιώ να παραιτηθεί. Και τώρα για το ΕΛΚ η κυρία Γκροστέφτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπω και πολλοί άλλοι θα απευθυνθώ στο Συμβούλιο. Διότι η σύνοδο αυτή είναι καθοριστική σημασία για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη, την ανάκαμψη τη οικονομία. Το ελπίζω να το γνωρίζουν τα κάτι μέλη, διότι οι ευρωπαϊκοί λαοί βαρέθηκαν να υποφέρουν δεν μπορούν πλέον να πιστέψουν στο μέλλον. Θα πρέπει να πω ωστόσο ότι η δήλωση του Συμβουλίου σήμερα μου φαίνεται πραγματικά ε, τελείω ε, δειλή και επιφυλακτική. Μα έχει συνηθίσει το Συμβούλιο βέβαια για να περνάμε από απογοήτευση σε απογοήτευση, αλλά δεν υπάρχει πια φιλοδοξία. Δεν υπάρχει δυναμικό χαρακτήρα για να προχωρήσουμε. Αυτό που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω απ' όλα δεν μπορούμε πλέον να καθυστερούμε και να χρονοτριβούμε. Ήρθε η στιγμή να περάσουμε στη δράση. Οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει επιτέλου να εκφράσουν πολιτική στήριξη ε, ισχυρή και άνευ ενδιασμών στο στρατηγικό πρόγραμμα επενδύσεων, στο πρόγραμμα παρουσίαση η Επιτροπή Juncker. Τα εργαλεία είναι στα χέρια μα. Εσεί πρέπει να τα πάρετε και να τα χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν συντομότερα. Και φτάνει, ε, α προσέχουμε τι χήμερε, διότι εάν δεν υπάρξει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, χωρί ε, οικονομική, δημοσιονομική και ε, σταθερότητα, χρηματοπροστατική σταθερότητα, δεν θα αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες. Χρειάζονται εδώ ιδιωτικέ επενδύσεις. Έτσι θα ε, στηριχθεί η πραγματική οικονομία. Και θα πρέπει ε, το ίδιο να γίνει και με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα ε, υπάρξει πραγματικά ανάπτυξη μόνο όταν τα κράτη-μέλη επιτέλους περάσουν στις ε, μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες Όσοι δεν λάβουν αυτή την απόφαση θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους λαούς τους. Είναι η στιγμή η Ευρώπη ε, να ε, ξεφύγει από την, ε, από την ανεξέλεγκτη δράση των εθνικών κυβερνήσεων. Είναι πολύ σημαντική η νέα προσέγγιση ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμά της. Λιγότερο γραφειοκρατική, περισσότερο στοχοθετημένη, πιο συγκεκριμένη. Τη συγχαίρω γι' αυτό και μόνο έτσι θα κερδίσουμε αυτή τη χρονική συγκυρία, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μα και με την Διατλαντική Συμφωνία εύχομαι πραγματικά η Ευρώπη να φανεί ισχυρή. Ισχυρή για να μην μείνουμε στο περιθώριο από τα νέα κέντρα τη Ασία και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τέλο, λίγα λόγια για ένα άλλο θέμα, την κατάσταση στην Ουκρανία. Ναι, είναι σοβαρή, ναι, πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία, αλλά είναι επίση πολύ σημαντικό να μην ακολουθήσουμε μία πολιτική, περιστική στην ε, πολιτική μας με αυτόν τον σημαντικότατο στρατηγικό εταίρο, τη Ρωσία. Και επίση να πω ότι δεν μπορούμε πλέον να αρκεστούμε στα, στα ημίμετρα. Πρέπει να υπάρξουν σαφή και φιλόδοξα συμπεράσματα. Και επαναλαμβάνω το τελικά λόγια του κυρίου Γιούγκερ. Θα ε, πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του επιτέλου στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής του Συμβουλίου, μια που παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου. Ο κύριος Γκερέρος Σαλόμ. Έλεγα ότι μια που είμαι εισηγητή για την ανθρωπιστική βοήθεια από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να πιστήσω την προσοχή σα σε ένα σημείο που πολλοί μπορεί να θεωρούν δευτερεύον και έχει να κάνει με το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αυτό είναι ο ιό του έμπολα. Δεν μπορεί να είναι περιθωριακό όμω ένα θέμα από το οποίο χάνουν τη ζωή του χιλιάδε άνθρωποι, ακόμα και αν βρίσκονται μακριά από εμά, μακριά από τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί πρέπει να στηρίξουμε την ε, απάντηση που δίνουμε. Εμείς, ναι, περιορίσαμε την ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ο ιός, αλλά δυστυχώς ο έμπολα εξακολουθεί να σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε το κοινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Και σε σχέση με τον κύριο Στυλιανίδη πρέπει να σας πω ότι πρέπει να στείλουμε γιατρούς, εργαστήρια, ιατρικές υπηρεσίες για να μην χαθούν τόσες ανθρώπινες ζωές και για να νιώσουμε μεγαλύτερη αξιοπρέπεια εμείς οι Ευρωπαίοι ανταποκρινόμενοι σε ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να βρίσκεται μακριά από τα σύνορά μας αλλά επηρεάζει τόσες ανθρώπινες ζωές. Ο Τούντα. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου επειδή υπήρξε τόσο μικρή στήριξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Ουκρανία. Δεν καλέθηκε ο κύριο Ποροσέγκο στην διάσκεψη κορυφή. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω το εξή. Εάν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι τέτοια που θα ζητήσετε και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, να συμμορφωθούν με τη συμφωνία του Μίνσκ. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση όσον αφορά και, τον και το θύμα και το θήτη τους βάζετε στην ίδια, σε δύο τσουβάλι. Δεν είναι σωστό όμως κάτι τέτοιο. Θέλω να πω λοιπόν τα Εμείς είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθούν στην ίδια κατάσταση όσον αφορά την κρίση μα. Σκεφτούμε τη συνοχή, σκεφτούμε τι χώρε οι οποίε μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004 και χρειάζονται συχνά πολύ περισσότερη στήριξη από τι χώρε οι οποίε βρίσκονται σε κρίση, επειδή η κατάσταση οικονομική αυτέ ήταν χειρότερη έτσι κι αλλιώ. Δυστυχώ όμω δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Ελπίζω να υπάρξει μια δίκαια κατανομή των πόρων. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Τελίτσκα, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπάμαι που ο κύριος συνάδελφος από το UKIP μετά από την καλλιτεχνική του παρουσίαση έφυγε. Γιατί θα ήθελα να του πω ότι γνωρίζω βρετανικές επιχειρήσεις που επενδύουν ε, και σε άλλες χώρες και ε, προσβλέπουν σε αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες που είναι και οι τρει πολύ σωστοί και πρέπει να εφαρμοστούν από κοινού. Και καλύτερε ρυθμιστικές διατάξεις το οποίο αναφερθήκατε, λαμβάνοντας υπόψη επίσης την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπέρ της οποίας είστε. Μία άλλη παρατήρηση. Σίγουρα το επενδυτικό σχέδιο θα μπορούσε να είναι πιο, πιο ολοκληρωμένο, να έχει λάβει υπόψη περισσότερο κάποιες προτάσεις της ομάδας μου. Έχω κάποιες αμφιβολίες για κάποια στοιχεία, αλλά είναι καλό επενδυτικό πρόγραμμα. Αυτό χρειάζεται η Ένωση, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις μας και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που πρότεινε η προηγούμενη Επιτροπή. Δεν με πείθουν βέβαια κάποια στοιχεία και δεν έλαβα απάντηση για την ανάγκη καλύτερου ρυθμιστικού πλαισίου. Ελπίζω να έχουμε μια ε, σταθερή βάση. Ωστόσο, προς το Συμβούλιο τώρα, κύριε Υπουργέ, η αρχική παρουσίασή σας με απογοήτευσε ιδιαίτερα. Με απογοήτευσε ιδιαίτερα. Ήταν πολύ γενικόλογη. Δεν αντιμετώπισε τα ουσιώδη θέματα. Σαν να μην έχει συνέστηση το Συμβούλιο του τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Ο κύριο Φερχόφστατ μίλησε για το πακέτο τηλεπικοινωνιών λέγοντας ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις αναμένουν και περιμένουν μήνες και χρόνια. Τι γίνεται για την ουδετερότητα του δικτύου, τι γίνεται για την περιαγωγή. Αυτά τα οποία προτείνεται είναι εντελώς ανεπαρκή. Κάτι άλλο με το οποίο καταλήγω δεν αναφέρθηκε. Το τέταρτο συνδρομικό πακέτο. Τι γίνεται με αυτό. Ούτε καν έχει ξεκινήσει και ήδη ε, ενώ μόλις έχει ξεκινήσει η συζήτηση λένε ότι θα διαχωριστεί το τεχνικό τμήμα. Όχι. Οι επιχειρήσει θα επενδύσουν μόνο αν σημειωθεί πρόοδο. Θα μπορούσα να αναφέρω και μια σειρά από άλλα θέματα. Δεν μα δίνεται ικανοποιητικέ απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ζητηθεί ε, μπλε κάρτα από τον κύριο Έθεριτζ. Το δέχεστε κύριε Στέριτσκα, ο κύριος Έθεριτζ. Ευχαριστώ που αναφέρθηκατε στην εξαιρετική ομιλία του συναδέλφου μου Πολ Νάταλ. Σίγουρα οι βρετανικέ επιχειρήσει θα έκαναν επενδύσει. Γιατί να μην επενδύσουν όταν υπάρχει περίπτωση να χάσουν. Αλλά δεν συμφωνείτε ότι ο λόγο που οι φορολογούμενοι πρέπει να φέρουν το κόστο αυτών των επενδύσεων είναι γιατί είναι κακέ επενδύσει. Είναι τόσο απλό. Αν δεν ήταν κακέ επενδύσει, οι ιδιωτικοί επενδυτέ δεν θα ήθελαν ε, κυβερνητική στήριξη μέσω χρημάτων φορολογουμένων. Ο κύριος Τερέτσκα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Σε ποιες επενδύσεις αναφέρεστε. Η απάντηση νομίζω είναι άλλη μια φορά απλή. Πιστεύω σταθερά στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά υπενθυμίζω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα που προτείνεται είναι να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις. Το ξαναλέω, μίλησα σε πολλούς Βρετανούς επενδυτές και θεωρούν ότι είναι πολύ καλό αυτό το πρόγραμμα Φυσικά μπορεί να έχουν κάποιες ε, παρατηρήσεις, αλλά είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση τους από αυτήν που ανέφερε πριν από λίγο ο συνάδελφός σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φορέντσα, επόμενος. Η κυρία Φορέντσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην προπαρασκευαστική συζήτηση θα θέλαμε από το Συμβουλίο να έχουμε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων τελείως διαφορετικό. Οι ζωές των πολιτών θα έπρεπε να βρίσκονται στο κέντρο των ανησυχιών σας. Αλλά ένα μόνο σημείο τους αφοσιώθηκε. Πώς θα ε, κατανείμετε τα εισοδήματα και την εργασία, πώς θα καλύψετε ε, ε, την έλλειψη ισορροπίας που έχουν δημιουργήσει πολιτικές λιτότητας. Αυτά θέλαμε να ακούσουμε. Από το Συμβούλιο αυτό θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη η έκθεση του ΑΣΕ που ε, μιλά για ανισότητες που εμποδίζουν την ανάπτυξη. όσα ε, δίνει μεγάλη έμφαση στην ανισότητα, την ανισότητα με απώλεια εισοδήματος που ε, έχει ε, συνέπεια για το ΑΕΠ 8,5%. Είναι τεράστιο αυτό το στοιχείο, αυτός ο αριθμός. Είναι τεράστιος και έχει χτυπήσει κυρίως τις ε, μέσες τάξεις και τις κατώτερες. Ε, έχει μακροοικονομικές συνέπειες. το εισόδημα λοιπόν θα πρέπει να μας αφορά ιδίω ως προς την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής, να επενδύσετε στην, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του πολίτε. Μιλάτε λοιπόν για σταθερότητα, αλλά τελικά στου ε, στους πολίτες την ανασφάλεια. Μιλάτε για εμπιστοσύνη, ενώ ο πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμπλέκεται σε ένα από τα σημαντικότερα σκάνδαλα με φοροδιαφυγή. Μιλάτε για επενδυτικό πρόγραμμα και ε, αυτό μοιάζει πάρα πολύ με τη μονόπολη που ξέρουμε ως επιτραπέζιο παιχνίδι. Ε, είναι σαν να δίνεται ελπίδε σε ένα άδειο κουτί και ελπίζουμε θα φτάσουμε τα 315 δις όταν στην πραγματικότητα στα χέρια μας έχουμε μόνο 21. Πείτε μου κάτι ε, για την Ιταλική Προεδρία στο εξάμεινο αυτό. Ο κύριος Ρέντσι συχνά λέει ότι σε αυτό το Ιταλικό εξάμεινο θα είχαν ε, αναλυφθεί μέτρα για την ανάπτυξη. Για το δικό σας εξάμεινο τι είδαμε, εκατομμύρια εργαζόμενοι να βγαίνουν στις πλατείες και να περνάνε σε γενική απεργία. Ευχαριστούμε ο κύριος Πρόεδρε, από τους διάφορους τομείς του δημόσιου βίου που χρειάζονται επένδυση επιγόντως, εγώ θα αναφέρω δύο που πιστεύω ότι έχουν μεγάλη σημασία. Επενδύσεις χρειάζονται στην έρευνα πρώτα απ' όλα που πρέπει να δούμε σε ένα πυλώνα πρόοδου και ευημερία στην Ευρώπη. Έρευνα σε όλους τους τομείς, στα πανεπιστήμια, στα μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα που δυστυχώς έχουν μειώσει πάρα πολύ τις δυνατότητες και πρέπει να ευνοήσουμε βέβαια και τη βιομηχανική έρευνα και την έρευνα όσον αφορά τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Και χρειάζονται επενδύσεις επίσης και στην πολιτική για την νεολαία, στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρθεση και στην απασχόληση. Κοινωνική και επιστημονική έρευνα στην πολιτική για τους νέους. Η έρευνα είναι το μέλλον και το μέλλον πρέπει να το προετοιμάσουμε ήδη από σήμερα διότι ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην κρίση είναι πολύ σημαντικό όπως σήμερα να φροντίσουμε το μέλλον. Είναι οι τομείς αυτοί, οι που πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαροί. Διαπιστώνω με μεγάλη έκπληξη ότι στην Ισπανία η κυβέρνηση, για παράδειγμα, περιορίζεται και μόνο μισή σελίδα έχει αναφέρει υπέρ τέτοιων επενδύσεων που όμως επιδέχεται ερμηνείες πολλές και διάφορες και τελικά καταλήγουμε σε αυθαιρεσίες. Επιμένω λοιπόν, χρειάζεται έρευνα και νεολαία. Αυτά τα δύο να φροντίσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Μόη, ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουν περάσει έξι μήνες από την ανάληψη της Προεδρίας από την Ιταλία. Έξι μήνες που τόσο πολύ περιμέναμε, δημιουργώντας προσδοκίες για τους πολίτες μας και την ανάπτυξη. Οπωσδήποτε η κυρία Μέρκελ ε, πρέπει να πούμε ότι έχει τις ευθύνες της όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως οι ιταλικές ευθύνες, οι ευθύνες της ιταλικής κυβέρνησης είναι προφανώς οι πιο σοβαρές, οι βαρύτερες. Η ιταλική κυβέρνηση λησμόνισε τελείω κάποιες προτεραιότητες και αφοσιώθηκε... Ε, ή για την ε, τόνωση τη αγορά εργασία ή για τη δημιουργία συνθήκων, δημιουργία θέσεων απασχόληση. Τέτοιε συνθήκε δεν θα δημιουργηθούν αν δεν επιλύσουμε κάποια κομβικά θέματα, ιδίω ό,τι αφορά τα θέματα τη μεταποιητική βιομηχανία. Είναι πολύ σημαντικό να, μειωθούν τα, να μειωθεί το κόστο για τι νέε και νεοφυεί επιχειρήσει. Να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Όταν μικρέ επιχειρήσει όμω και βιοτεχνίε κλείνουν, πώ θα γίνει αυτό. Ε, είναι πολύ ε, είναι υπερβολική και περιττή γραφειοκρατία που ε, σφίγγει σαν μέγενη την Ιταλία και την Ευρώπη. Η Ιταλική κυβέρνηση ε, είχε υποσχεθεί αγώνα για το Made in, για να υπάρξει ε, νέα ε, δραστηριότητα στην, στις επιχειρήσεις της Ευρώπης και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έπρεπε να καταπολεμήσει την πειρατεία και την παραποίηση με ένα κοινό τελωνιακό σύστημα και μια ελεύθερη αγορά όπως στην Ευρώπη θα έπρεπε να ελπίζουμε ότι θα γίνει. το για την προστασία των επιχειρήσεων. Δεν έγινε τίποτε. Τίποτε δεν έγινε επίση για να αντιμετωπίσουμε τη διάσωση των μεταναστών. Ε, για να μην πούμε ότι επί 40 χρόνια ε, ε, κλέψατε κονδύλια που, έπρεπε να κατευθυνθούν αλλού. Το ίδιο και από του μετανάστε, όπω μάθαμε στο σκάνδαλο προχθέ. εκατομμύρια κλέψατε από αυτού του καημένου, που εκατομμύρια που θα έπρεπε να έχουν στηρίξει την Ιταλία και την Ευρώπη. Η Προεδρία σας έπρεπε να έχει εντείνει τον έλεγχο, δεν το έκανε και μάλιστα αποσιώπησε το όλο πρόβλημα. Αυτά ήταν τα κατεπήγοντα θέματα που έπρεπε να έχει αναλάβει η Ιταλική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αν ε, ε ήθελε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να συντονιστούν. Τώρα φαίνεται να συμμετέχουν όλοι σε έναν οργανισμό τύπου μαφίας και αυτό είναι μια ντροπή. Πώς να υπάρξουν δουλειές αν δημιουργήσετε θέσεις εργασίας. Πώς ε, θα υπάρξει πολιτική εάν κλέβατε χρήματα τόσα χρόνια. Είσαστε όνειδος. Uh, Υπάρχει μία μπλε κάρτα. Τη δέχεστε παρακαλώ. Η, η κυρία Ρεσόβα. Ε, Βρέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω την ε, συνάδελφο εάν νομίζει ότι είναι στην Ιταλική Βουλή ή αν γνωρίζει ότι βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ μιλούμε για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επ' αυτού δεν μας είπε απολύτω τίποτε και νομίζω ότι η Ιταλική Προεδρία ήταν εξαιρετική μαζί με όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι η τη ενώση, εάν χάναμε όλοι μαζί ψηφίζαμε όλοι μαζί, εκεί θα κρινόταν το αποτέλεσμα. Και βεβαίω ε, ε, για το πρόγραμμα εργασία το οποίο συζητάμε, ε, θα πω και εγώ τη γνώμη μου, αλλά η συνάδελφο δεν είπε τίποτε, τίποτε και αυτό ακριβώ είναι το θέμα μα αυτή τη στιγμή. Ε, κυρία Μόε, η Ιταλία ε, ζει σε διαφορά. Συνεχώ αποκαλύπτονται σκάνδαλα. Στη Ρώμη η μαφία είναι ανεξέλεγκτη. Έχουν κλαπεί κονδύλια από παντού. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα και δεν ζητήσουμε βοήθεια από την Ευρώπη, πώ θα ε, σωθούμε. Η Ιταλία πτωχεύει, είναι σε default. Εάν δεν προχωρήσει η Ιταλία, δεν θα προχωρήσει ούτε και η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κόρβιν μέχρι για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν κάτι πολύ απλό. Για να καταπολεμήσουμε την ανεργία χρειάζονται χρήματα. Και για να βρουν χρήματα φορολογούν. Δημιουργούν λοιπόν θέσει εργασία με τα χρήματα και τι χάνουν μέσω τη ε, αύξηση των φόρων. Τόσο απλό είναι. Ε, μια εταιρεία φοροδιαφεύγει, παράγει φτηνότερα πουλάει περισσότερα. Αν πουλάει περισσότερα, δημιουργεί θέσει εργασία. Χάρη στον κύριο Γιούνκερ, ω πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, όχι χάρη στον κύριο Γιούνκερ, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταργηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γκαρντίνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα Κάνουμε νομίζω μια συζήτηση ζωτική σημασίας. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία με το Συμβούλιο αυτό που εντός λίγων ημερών θα διεξαχθεί να συζητήσουμε κι εμείς πράγματα που μας απασχόλησαν και στο εσωτερικό του ΕΛΚ. Να θυμίσω τα έγγραφα του συνόδου που οργανώσαμε στο Δουβλίνο, της διάσκεψης την περασμένη άνοιξη και επιτέλους μπορούμε να δώσουμε σάρκα και οστά αυτά που είπαμε, στα λόγια μας. Αλλά τώρα επιτέλους πρέπει να δράσουμε. Απευθύνομαι λοιπόν στον πρόεδρο Γιούνκερ, ε, που έχει, στον οποίο εμπιστευθήκαμε τις ελπίδες μας και ελπίζω να δώσει την ευκαιρία σε αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα να γίνει ε, μία ευκαιρία ώστε να διορθωθούν ανισορροπίες ε, και ανισότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Όλα αυτά είναι θέματα που αν δεν τα αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο θα εκμηδενήσουν και θα αποδυναμώσουν την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού προγράμματος. Το χρειαζόμαστε όμως το πρόγραμμα αυτό, διότι μας λέγατε πρόσφατα ότι 100 ε, δις έχουν ήδη φύγει προ το εξωτερικό. Δεν είναι ελκυστικέ οι χώρε μα για τι επενδύσει. Αυτό νομίζω είναι το πλέον καθοριστικό θέμα που πρέπει να μελετήσουμε. Επίση, το θέμα των πλεονασμάτων, πλεονάσματα δύο χωρών τη Ευρωπαϊ... της Αυτό πρέπει να το δούμε κατά πρόσωπο, διότι από την άλλη όχθη του Ατλαντικού μα ρωτούν τι κάνουμε οι Αμερικανοί. Και εδώ, Πρόεδρε, Σα ρωτώ, δεν πρέπει να εξετάσετε και αυτό το στοιχείο το εμπορικό του πλεονάσματος ουσιαστικά δημιουργεί ενδιασμού στους Αμερικάνους για να προχωρήσουν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην συμφωνία, την συμφωνία, το TTIP, διότι ακόμη οι Αμερικανοί δεν έχουν συμφωνήσει στην απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει προτεραιότητά τους το TTIP. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί επικεντρώνονται ε, ως επιτοπλίστων την διατλαντική εταιρική σχέση. Σε αυτές τις ερωτήσεις λοιπόν ελπίζω να μου δώσετε απάντηση και να ευχηθώ καλή δουλειά στο Συμβούλιο, ελπίζω, ελπίζοντας ότι θα αντιμετωπίσει την έλλειψη εμπιστοσύνη των ε, πολιτών και θα την καλύψει όλα τα κενά. Ευχαριστούμε, κυρία Κέπχαρτ. Ευχαριστώ. Και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω έκκληση προς το Συμβούλιο πολύ σημαντική έκκληση να συμβάλλει το Συμβούλιο ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Είναι πολύ ουσιώδες αυτό. Αλλά να μην ξεχάσουμε και το εξή. Στο κέντρο της προσοχής μας δεν πρέπει να είναι μόνο η ανάπτυξη γενικά, γενικόλογα. Πρέπει να έχουμε υψηλή αξία και βιώσιμες θέσεις εργασίας και βιωσιμότητα γενικότερα. Αυτό σημαίνει όμως να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και αυτό δεν το βλέπω στην ουσία ε, ο καθένας προτείνει κάτι το δικό του ποτίζουμε λίγο εδώ λίγο εκεί όχι πρέπει να επικεντρώσουμε να εστιάσουμε στα σημαντικά καθήκοντα στους καινοτόπους τομείς που θα δημιουργήσουν υψηλού επίπεδου θέσεις εργασίας για παράδειγμα ψηφιακό θεματολόγιο βιωσιμότητα στον ενεργειακό τομέα υποδομές ούτως ώστε πραγματικά να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεμές Μάκερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω λιγάκι στην κατάσταση στην Ουκρανία. Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεσμεύεται να προχωρήσει με τη Συμφωνία Σύνδεσης. Αυτό είναι θετικό. Είναι θετικό όλες οι χώρες μέλη να αποφασίσουν και να συμφωνήσουν την επικύρωση μια τέτοια συμφωνίας. Η κυριαρχία της χώρας είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και οι μεταρρυθμίσεις βέβαια που έχουν ζητήσει σαφώς οι πολίτες της Ουκρανίας. Η Ουκρανία βέβαια για να το πετύχει αυτό χρειάζεται τη βοήθειά μας. Στο μεταξύ βλέπουμε ότι οι κυρώσεις κατά του Πούτιν έχουν κάποια αποτελέσματα. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να ε, φυσικαστούμε. Το θέμα της παράνομης προσάρτησης είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσει να μας απασχολεί. Σε ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, Κρυμαία, συζητήθηκε και το θέμα των ρωσικών διαβατηρίων που δίνονται στους κατοίκους της Κρυμαίας. Θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τα διαβατήρια αυτά είναι σαν έμεσα να αναγνωρίζουμε την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Πρόεδρος, έχετε... Κύριος Λάμπστορ, μάλλον τώρα. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, Θέλουμε την επιτυχία τη Ένωση, θέλουμε την επιτυχία αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρία στοιχεία είναι αποφασιστικά. Ένα καλό πρόγραμμα εργασιών, κύριε Γιούγκερ, Το πρόγραμμά σα είναι πολύ καλό. Είχατε το θάρρο ε, να αλλάξετε άποψη, να αλλάξετε προσέγγιση με τη βοήθεια και του κύριου Τίμερα, μα από ό,τι φαίνεται, και να στραφείτε προ νέου τομεί. Δεύτερον, που βλέπουμε από το πρόγραμμα τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαρθρωτικέ αλλαγέ στα κρατη Έχουν πολλέ ανησυχίε στην Ιταλία, στη Γαλλία και στο Βέλγιο που επιχείρησε για παράδειγμα να κάνει μετροπαθείς μεταρρυθμίσεις είδαμε γενική απεργία τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξα αν θέλουμε να καταλήξουμε σε επιτυχία και τρίτον πρόγραμμα επενδύσεων από πολλούς επικρίνεται νομίζω ότι είναι λάθος λάθος ήδη ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ότι οι κρατικές εγγύησεις ε, δεν θα βοηθήσουν στο παρελθόν βοήθησαν γιατί να μην βοηθήσουν και τώρα αυτό θα επιδιώξουμε ένα είναι σημαντικό Είπατε ότι θα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα προγράμματα. Αυτό είπατε την προηγούμενη φορά. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό. Να μην κάνετε όμως το λάθος να πιέζουν τα κράτη-μέλη για τα προγράμματά τους. Η γερμανική κυβέρνηση ζήτησε να επιδοτηθεί η δημιουργία του, του αεροδρομίου Βερολίνο-Μπράντεμπουργκ, το οποίο είναι ήδη αποτυχία. Μην επιδοτήσετε τέτοιο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λάμπτορφ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Παπαδημούλης. Το νεοφιλελεύθερο δόγμα ότι η μονομερής λιτότητα θα αυξήσει τις επενδύσεις δοκιμάζεται κύριοι του Συμβουλίου και της Κομισιόν έξι χρόνια τώρα και οι επενδύσεις έχουν μειωθεί κατά 15% άρα χρειάζεται μια στροφή στην πολιτική με περισσότερους δημόσιους πόρους για την ανάπτυξη και από τον κοινωνικό προϋπολογισμό και από τα κράτη μέλη. κύριε Γιούνκερ, το πακέτο που μας παρουσιάσατε είναι σχεδόν άδειο γιατί μόνο ο ιησούς χριστός πολλαπλασίασε τα ψάρια και τα ψωμιά με το γνωστό θαύμα. μόχλευση με αυτές τις συνθήκες οικονομίας 1 προς 15 είναι αδύνατο να επιτευχθεί και σας το λένε σχεδόν όλοι. Αλλά κύριε Ντελαβέντοβα, εσείς στο σχεδόν άδειο πακέτο του κυρίου Γιούνκερ προσπαθείτε με την αναβλητικότητα και τα ευχολόγια να το αδειάσετε εντελώς. Ποια θα είναι η συμμετοχή των κρατών μελών, με ποια κριτήρια, πώς διασφαλίζετε ότι οι επενδύσεις θα εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη και θα ενισχύσουν τη συνοχή. Για όλα αυτά δεν μας λέτε τίποτα και πολύ φοβάμαι ότι το Συμβούλιο Κορυφής θα οδηγήσει απλώς σε χριστουγεννιάτικες ευχές. Ευχαριστώ πολύ. Η Μισόλ Ριβαζή, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να λάβω το λόγο για την επιδημία έμπολα και για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει για το σημαντικό αυτό φαινόμενο. Οι ειδικοί λένε ότι έχει να κάνει με την αποψήλωση των δασών, με το σύστημα υγειονομική περίθαλψη και την πολιτική αστάθεια τη εν λόγω περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιέρωσε 1,1 δι ευρώ ανθρωπιστική βοήθεια για την καταπολέμηση του έμπολα και 440 περίπου ευρώ προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περίεργο αλλά συνέβη. Το πρόβλημα είναι ότι οι υπουργοί αύριο συγκεντρώνονται για να υπογράψουν, υπέγραψαν στις 12 ε, Δεκεμβρίου την ίδια χρονιά την ε, Συμφωνία Εταιρική Σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Περίεργο και αυτό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε εμπορικέ ε, προτιμήσει μονομερεί στι πρώην απικίε τη στι εταίρου και ακόμη με του δασμούς δασμού παίρνει αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τα πληρώνει με το σύστημα που έχει προβλέψει. Κατάργηση των δασμών για το 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Αυτό συνέβη. Χρειάζονται όμως κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές τους και δεν τα λαμβάνουν πλέον με τους του τους δασμούς. Τι θα κάνουν αυτές οι χώρες. Πέτερ δύο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ο κύριος Γιούνκερ λέει ότι χρειάζεται περισσότερα χρήματα. Δεν με εκπλήσει γιατί ότι να έχει κανείς την ευθύνη για τα χρήματα των φορολογούμενων είναι κάτι το οποίο σπάνια βλέπουμε εδώ σε αυτό το σώμα. Αν δείτε την κατάσταση που επικρατεί εδώ σε σχέση με την οικονομική κατάσταση που έχουν οι άνθρωποι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε πρώτα απ' όλα ότι το 43% των πολιτών αποφάσισαν να μην ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. 30.000 ευρώ δίνονται σε ε, αμοιβέ για αυτούς οι οποίοι φεύγουν από το αξίωμά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρήματα πληρώνονται λοιπόν ενώ η φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο χαμηλή από εκείνη που έχουμε για παράδειγμα στο Βέλιο. Αν λοιπόν παίρνετε χρήματα όταν τελειώνετε την απασχόλησή σας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράλογο. Γιατί να δίνονται αυτές οι αμοιβέ. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα μπόνους δηλαδή. Ενώ οι άνθρωποι εκτός ε, θεσμικών οργάνων στην Ευρώπη μόνο πληρώνουν, πληρώνουν και ξαναπληρώνουν. Ο κύριος Γιούνκερ λέει ότι θέλει να επανακτεθεί εμπιστοσύνη. Πώς θα γίνει αυτό. Δείτε πώς διαχειρίζεται το σώμα αυτό τα χρήματα των φορολογούμενων. Είναι μια αδύνατη αποστολή αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για την ίδια τους την ύπαρξη. Πώς είναι δυνατόν να έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι αυτοί σε αυτά τα οποία βλέπουν να συμβαίνουν εδώ. Η κυρία Μπιτσότο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα έχει όλο και το... θα έχει όλο νέα, ε, νέα εκτελεστική εξουσία και νέο Πρόεδρο. Πολλά ακούσαμε λοιπόν, πολλά λόγια, αλλά δεν βλέπουμε καμία τολμηρή επιλογή. Δεν θα αλλάξει τίποτα για του πολίτε, για του ανέργου, τη επιχειρήση. Για του ανέργου που μένουν χωρί μέλλον, ε, με άδεια τα χέρια. Μόνο επιουσχέσει έχουμε ακούσει. Ε, βλέπουμε να μένουμε πάντοτε στα ωραία λόγια πώς ε, διαγράφεται το τέλος του 2014, το τέλος του εξαμήνου της Ιταλικής Προεδρίας, με τόσα άδεια και ωραία λόγια, όπου ακούσαμε τους πρόεδρους Ρέντζι να μας, κάνει, να μας δίνει πολύ ε, υποσχέσεις, τις οποίες επικροτήσαμε πριν από πολλούς μήνες, αλλά πείτε μου, ένα πράγμα έγινε κάτι θετικό για τους Ιταλούς πολίτες και τους Ευρωπαίους πολίτες από την Προεδρία του Ρέντζι. Μας υποσχέθηκε να αλλάξει την Ευρώπη. Τον Μάιο, λίγου μέρε πριν τι ευρωεκλογέ. μας είπα ότι θέλω μια Ευρώπη ανθρώπινη, μια Ευρώπη που να μην ασχολείται πώ θα σώσει τι ε, ε, τράπεζε, αλλά τι οικογένειε. Αυτά μα είπε και ο κύριο Γιούγκερ, πρόεδρο τη Επιτροπή. Ευχαριστούμε, Ματέο Ρέντσι, αλλά ήταν γελία όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εστέβαν Γονθάλεφ Πόνς, ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Γιούγκερ. είναι πολύ σημαντικό το επόμενο συμβούλιο και εγώ θα σα μεταφέρω τι περιμένουν από το Συμβούλιο αυτό οι ψηφοφόροι μου που σας στηρίζουν. Θέλουν συντονισμό προκειμένου να ευνοηθούν οι επενδύσεις και να ενισχυθεί μια αγορά. Θέλουν επίσης να ενισχυθεί ο αγώνας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι Ισπανοί πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για μια πραγματική ενεργειακή ένωση στην Ευρώπη, να έχουμε ανταγωνιστική αγορά με τις διασυνδέσεις που χρειάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ενέργεια σε ικανοποιητικές τιμές. Θέλουν επίσης στην Ευρώπη να είναι ένας ασφαλής χώρος. πολέμηση της τρομοκρατίας, να λυθεί το πρόβλημα αυτό από την επιστροφή των ξένων μαχητών να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους στόχους μας. Κύριε Πρόεδρε, είναι βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει μετά από τη δολοφονία πάνω από 100 παιδιών στο Πακιστάν. Κάθε φορά που χάνει τη ζωή του ένα παιδί σε ένα σχολείο είναι σαν να χάνει τη ζωή του ένα παιδί στο σχολείο της Ευρώπης. Το πνεύμα της Μαλάλα πρέπει να μας συνοδεύσει στον αγώνα μας αυτό κατά της τρομοκρατίας. Έπειτα, χρειάζεται αλληλεγγύη για να είναι πραγματικότητα τα κοινά μας σύνορα. Τώρα που δεν έχουμε εσωτερικά σύνορα, πρέπει να πω ότι με λίγια η Θέουτα αποτελούν επίσης σύνορα και της Γαλλίας και της Σουηδίας και όλων των ευρωπαϊκών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε για την Ουκρανία αλλά και για τη Ρωσία. Πρέπει να προβλέψουμε τι συνέπειες θα είχε για την οικονομία μας, για την απασχόληση στην Ευρώπη, η κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας αν αυτό συμβεί τον επόμενο χειμώνα. Τα χθεσινά νέα και σημερινές ειδήσει πρέπει να μας ανησυχήσουν, να μας απασχολήσουν οι ψηφοφόροι μου λοιπόν ζητούν μετά το Συμβούλιο, όταν θα έχει τελειώσει αυτό, να αρχίσετε τις εργασίες σας με κάθε επιτυχία. Κύριε Γονθάλεθ Πόντς, ο κύριος Τέρη Κάμπρας ε, έχει ζητήσει μια μπλε κάρτα. Κύριε Τέρη Κάμπρας, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Είναι πολύ καλό αυτό που λέτε για την ενέργεια στην Ευρώπη. Πώς εξηγείτε ότι η ενέργεια στην Ισπανία είναι πιο ακριβή από ό,τι σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί προστατεύεται η ευρωπαϊκή ενέργεια, γιατί δίνουμε δώρα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, μάλλον ένα δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια ευρώ τα χαρίζουμε. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα χρήματα αυτά πληρώθηκαν σε πολύ μέσα σε 30 μέρες. Γιατί λοιπόν μιλάτε για την ευρωπαϊκή ενέργεια χωρίς προηγουμένως να έχετε τακτοποιήσει τα όσα συμβαίνουν στην Ισπανία με την τιμή της ενέργειας. Ο κύριος Τερκάμπρα μου μιλάει στα ισπανικά σε αυτό το σώμα, το απαντήσω κι εγώ. Κοιτάξτε, η Ισπανία προσπαθεί να μειώσει το κόστος της ε, ενέργειας για τους Ισπανούς, αλλά θέλει επίσης η ενέργεια να είναι ανταγωνιστική και να αποτελεί ένα μέσο πρόοδο για την Ισπανία και για την Ευρώπη. Πολύ θα θέλαμε η Ιβηρική να ενωθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω των Πυρηναίων, ώστε το φυσικό αέριο από την Αλγερία να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να υπάρξουν προβλήματα με το ρωσικό τον επόμενο χειμώνα. Υπάρχει και δεύτερη μπλε κάρτα τον κύριο Σαν, δέχεστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αναφέρατε στην ομιλία σας ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροποφυγής. Το κόμμα σας θα ήταν αποφασισμένο δηλαδή να τα βάλει με χώρες οι οποίες επιβάλλουν υπερβολικά πολλούς φόρους στους πολίτες. Και το αποτέλεσμα είναι να ενισχύεται η μαύρη οικονομία όπως συμβαίνει στην Ουγγαρία. Απάντηση. Ναι. Η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Περβάνς Μπερές. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στην Ιταλική Προεδρία γιατί θα πρέπει να κινητοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί για την ψηφιακή οικονομία. Ο καθένα φαντάζεται ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που θα απασχολήσουν και το επενδυτικό πρόγραμμα και θα ε, δημιουργηθεί από αυτό κέρδο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τουλάχιστον ανακοινωθεί και εκφράζουμε την ικανοποίησή μα όμω. Μόνον αυτή η καρπή των επενδύσεων ε, επιστρέψεων στα χέρια των Ευρωπαίων θα έχει νόημα όλη αυτή η προσπάθεια. Οι ψηφιακέ επενδύσει λοιπόν και η φορολογία είναι ένα σημαντικό ε, θέμα. Εκεί θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορούμε να πάρουμε ε, ένα ε, μέρος του κέρδους από τις εταιρείε θα πρέπει να το θέσετε στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το ίδιο και την προστασία των δεδομένων. Ιδάλλως θα έχουμε διαφυγή τις γνώσεις και των κεφαλαίων που δεν θα καταφέρουμε να κρατήσουμε εδώ. Και να απευθυνθώ και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι σε αυτό το Συμβούλιο θα προσπαθήσετε να καθορίσετε ένα φύλλο πορείας για το μέλλον της Ευρωζώνης. Όταν ακούω όμως τον κύριο Βέμπερ, ε, ε, ανησυχώ κάπως, διότι δεν νομίζω ότι στυλιτεύοντας ε, ή προσβάλλοντας ε, μεν τους δε θα μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο στην Ευρωζώνη. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι να ε, αποδεχτούμε τις αλληλεξαρτήσεις μας και την αλληλεγγύη μας για να μας αναγνωρίσει και ο υπόλοιπος κόσμος μία, ε, ως μία δύναμη αναδεικνύοντα την κοινή μα δύναμη να ανταποκριθούμε σε απαιτήσει που σήμερα, συνάδελφοι, έχει ολοκληρωθεί ο χρόνο σα, Ολοκληρώνω τη φράση μου. Ε, δεν μπορεί να διορθωθούν λοιπόν οι ανισότητε με τα εργαλεία που αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και τώρα δεν θα χορηγήσω μπλε κάρτα, δεν θα επιτρέψω μπλε κάρτα, διότι υπερεύει το χρόνο της η κυρία Μπερέζ. Ο κύριος Μπέρντ και ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, Ακούσαμε μια αξιοπρόσεκτη ομιλία του επικεφαλής των φιλελευθέρων, κύριο Φερχόφστατ. Ο κύριος Φερχόφστατ θα παρατήρησε, ελπίζω να έχει παρατηρήσει, ότι η Ευρωζώνη είναι σε μια πολύ σοβαρή και βαριά κρίση. Το είπε ο ίδιος. Τι σημαίνει αυτό για ένα πρόεδρο φιλελεύθερης ομάδας που συνήθως ε, φοράει ροζ γυαλιά όταν μιλάει για την Ευρώπη. Για πρώτη φορά ε, επικρίνει το Συμβούλιο γιατί δεν προτείνει λύσεις. Αυτή είναι λάθος ανάλυση. Το Συμβούλιο πρέπει να μας κάνει σωστή ανάλυση. Γιατί έχει προκύψει αυτή η κρίση. Γιατί αυξάνεται η οικονομία στην ε, Νότια και Βόρεια Αμερική, γιατί στην Αποανατολή, γιατί στην Οκεανία, ε, την Αυστραλία, γιατί οι χώρες εκτός της Ευρωζώνης στην Ευρώπη παρουσιάζουν ανάπτυξη, αλλά όχι Ευρωζώνη. Και γι' αυτό σα ρωτώ, κύριε εκπρόσωπο του Συμβουλίου, γιατί δεν έχουμε οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, γιατί έχουμε αυτή την περίφημη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κοινό νόμισμα, την ενιαία αγορά, γιατί όμω δεν έχουμε ανάπτυξη. Γιατί, σα παρακαλώ να το σκεφτείτε σοβαρά. Κύριε Λούκε, ο κύριο Λάμπτορφ θέλει να σα κάνει μια ερώτηση με μπλε κάρτα, το δέχεστε. Παρακαλώ κύριε Λάμπτορφ, 30 δευτερόλεπτα. Δύο ερωτήσει προ τον Σάλφο Λούκα. Η πρώτη έχει υπόψη του ότι οι δραστηριοτικέ μεταρρυθμίσει σε σοβαρά κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη δεν έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει επαρκώ, ούτω ώστε να υπάρχει πραγματικά ανάπτυξη. Γαλλία και Ιταλία, τι ανέφερα ήδη στην ομιλία μου. Η Γαλλία μα προκαλεί τι περισσότερε ανησυχίε. Δεύτερη ερώτηση. Πότε για τελευταία φορά ήταν τόσο κοντά στον ε, Γκί ε, Φερχόφστατ ώστε να διαπιστώσει ότι φοράει ροζ γυαλιά. Λούκε. Κοιτάξτε, έχω πολύ καλή όραση και βλέπω και από τόσο μακριά. Όσον αφορά τι διαστοτικέ μεταρρυθμίσει, έχετε δίκιο. Δεν έχουν γίνει οι διαστοτικέ μεταρρυθμίσει. Και γιατί δεν έγιναν. Αυτό οφείλεται στο ότι εσεί και οι φίλοι σας ακύρωσαν τη ρήτρα μη κοινή ανάληψη ευθυνών για τα χρέη. Εάν δεν είχε ακυρωθεί αυτή η ρήτρα, οι κράτες, οι, τα κράτη-μέλη θα είχαν ε, εφαρμόσει πολύ σοβαρότερε μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Από εδώ και στο εξή θα τηρώ αυστηρά το χρόνο για να μπορούν να γίνουν περισσότερες ερωτήσεις μέσω μπλε κάρτας, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Σας παρακαλώ λοιπόν να τηρείτε επακριβώς το χρόνο σας. Ο κύριο Όλη Ρέν ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη χρειάζεται την ανάπτυξη και την απασχόληση και απαιτούνται επενδύσεις, ιδίω ιδιωτικές. Υπ' αυτήν την έννοια, το επενδυτικό πρόγραμμα του κυρίου Γιούνκερ είναι αξιέπαινο. Η Ευρώπη πρέπει να μεταρρυθμιστεί ώστε να προσελκύσει επιτέλους επενδυτές με ένα καλό κλίμα για τις επενδύσεις, με την ενιαία αγορά να λειτουργεί για την ψηφιακή οικονομία και τις υπηρεσίες, με μια εσωτερική αγορά που αυτή τη στιγμή έχει πολλά κενά και που θα πρέπει να καλυφθούν με, αρκτικές, με επενδύσεις που θα πρέπει να οδεύσουν, να οδεύσουν προς την Αρκτική και τόσες άλλες προτεραιότητες με διευθυντικές μεταρρυθμίσεις σε μεγάλα κράτη όπως η Γαλλία και η Ιταλία η ανάπτυξη πρέπει να ε, προχωρήσει και μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως η Γερμανία ε, που αξιοποιεί το περιθώριό της ε, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το ίδιο και η ΕΚΤ, αν όχι από τα Χριστούγεννα, από το νέο έτος. υπάρχει η γαλάζια κάρτα από τον κύριο Παπαδημούλη, τα 30 δευτερόλεπτα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρεν, αυτές τις μέρες αναπτύστε μια κινδυνολογία και μια προπαγάνδα ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις πιθανότατα επερχόμενες εκλογές στην Ελλάδα θα σημαίνει την έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ και μια μεγάλη καταστροφή για την ίδια την ευρωζώνη. Πώς σχολιάζετε αυτή την εκστρατεία φόβου. Okay. Ευχαριστώ κύριε Παπαδημούλη. Η Ελλάδα είχε κάποιε δυσκολίε στο παρελθόν, τώρα πάλι αυτέ αυξάνονται. Δεν έχω καμία διάθεση παρέμβαση στη εσωτερική σα πολιτική και στα εσωτερικά πολιτικά σα πράγματα. Όμω καταλαβαίνω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο Τσίπρα είναι δεσμευμένη ε, ως προς την συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αυτό νομίζω ότι μετράει και αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Επίσης κατανοώ ότι είναι πολύ βαρύ το βάρος του χρέους. Θα πρέπει να προχωρήσει λοιπόν σε μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα. Κοιτάζοντας τι θα γίνει και με τα δάνεια που προχωρούν, όχι αναγκαστικά αντλώντας από κεφάλαια. Ο κύριος Μπίτικοφ, ένα λεπτό, ευχαριστώ. Ο κύριε Πρόεδρε Γιούγκερ, ε, κυρίες και κύριοι, στην αντιπαράθεση για το πώς θα αποτελέσει μια νέα έναρξη για μόνιμη ανάπτυξη το πρόγραμμα Juncker, το πρόγραμμα επενδύσεων Juncker, εμείς ως πράσινοι απαιτούμε πάνω απ' όλα όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλουν με δικούς τους πόρους σε αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα. Παρακαλώ τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, αυτό που όλες οι πλευρές του σώματός μας το έχουν διατυπώσει, να το λάβει σοβαρά. Δεύτερον, όσον αφορά τα ίδια τα προγράμματα που πρέπει να εφαρμοστούν, υπάρχουν έξι ουσιώδη κριτήρια. Πρώτον, όπως είπε ο κ. Γιούνκερ, δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, κλαδικές ή γεωγραφικές ποσοστώσεις. Πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πρέπει να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να επιλέγονται μέσω εμπειρογνωμόνων της Τράπεζας Επενδύσεων με, που να έχουν γνώση των θεμάτων. Πρέπει να συμμετέχουν ιδιωτικές επενδύσεις και να προωθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαριανόπουλος. Ένα λεπτό. Σύνοδος κορυφής θα κλιμακώσει την αντιλαϊκή επίθεση. Όπως τις επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και αλλού, που θα φέρουν νέα κύματα προσφύγων. ενισχύεται η απειλή γενικευμένου πολέμου στο βωμό ανταγωνισμών για νέες αγορές στην ενέργεια και τους δρόμους μεταφοράς της. ομολογείται ότι την ασθενική ανάκαμψη μπορεί να ακολουθήσει νέα οικονομική κρίση που δεν μπορούν να σταματήσουν ούτε οι υπερασπιστές της περιοριστικής πολιτικής ούτε της χαλάρωσης που ομοφωνούν όμως μεταξύ τους για πάνθινη δουλειά κατεδάφιση δικαιωμάτων ξερίζωμα της αγροτιάς αντιλαϊκούς φόρους επιβάλλονται τα μόνιμα μνημόνια με καταστολή των αγώνων. φορτώνονται οι λαοί με χρέη που δεν οφείλουν αφού το κρατικό χρήμα όπως τα 300 δις του πακέτου Γιούγκερ, πηγαίνει στις επιχειρήσεις. οι ανταγωνισμοί επιχειρηματικών ομίλων κυβερνήσεων και κομμάτων που τους εκπροσωπούν δεν αφορούν τα λαϊκά συμφέροντα. η ευρωπαϊκή ένωση δεν γίνεται φιλολαϊκή. είναι ώρα ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής και να ανατρέψει αυτή τη βαρβαρότητα. Ευχαριστώ πολύ. Άντρα Κιούρκ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αξιότιμοι συνάδελφοι, προκειμένου να μας η ευρωπαϊκή οικονομία, κάτι με το οποίο όλοι συμφωνούμε και συμφωνώ και εγώ με τους στόχους, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, γι' αυτό και έχω να κάνω τα σχόλια πέρα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν υπάρχει φρέσκο χρήμα, νέο χρήμα. Και αν δείτε τον ορίζοντα 2020 ή το συνδέοντα στην Ευρώπη, πολλά πράγματα δεν υπάρχουν. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι βγάζουμε τα χρήματα από τη μια τσέπη και τα βάζουμε στην άλλη. Και αν δείτε και το πολυπλασιαστικό φαινόμενο, τη μόχλευση, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ αισιόδοξη. Αν δείτε τις εκτιμήσει, εγώ δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικέ. Δυστυχώς. Έπειτα, λαμβάνοντας υπόψη μας την ε, συνένεση που θέλουμε, πρέπει να συμφωνήσουμε και με τα προγράμματα, γιατί μόνο προγράμματα πραγματικά ποιότητας μπορούν να βοηθήσουν να έχουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα που τελικά θα στηρίξουμε θα είναι ικανοποιητικά και θα συνάδουν με τους στόχους μας. Κάποια προγράμματα όντως συνάδουν με τους στόχους μας το θέμα της ασφάλειας ενέργειας. Όμως, την ενεργειακή διάσταση την είχε τονίσει και η Επιτροπή Παρόσο. Εμείς πρέπει να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα λέμε ότι έχουμε πόρους για πράγματα για τα οποία δεν έχουμε. Έχουμε ένα μεγάλο και σημαντικό ρόλο να παίξουμε. Θέλουμε τιμές ενέργειας που να μπορούν να πληρώσουν οι πολίτες. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να έχουμε μια πραγματικά ενέργειακή αγορά. Η φτηνή ενέργεια θα βοηθήσει την Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ. Μπλε κάρτα από το κύριο Γιουλελή. 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή. Προκειμένου η οικονομία να μπει και πάλι στο αυλάκι και να ανακτηθεί εμπιστοσύνη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως Ούγγρος βλέπω ότι για κάποιες χώρες, όχι μόνο για τη δικιά μου, υπάρχουν πολιτικά κόμματα όπου ο Πρωθυπουργό όπως ο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας τα λέει αλλιώ τα πράγματα για την Ευρώπη. Εσείς τι έχετε να πείτε για το νέο φόρο, για παράδειγμα, που έχει εισαχθεί και για το ότι ο Πρωθυπουργό τα βάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι εκείνη φταίνει, εμεί ξέρουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Τι λέτε για αυτήν την ε, άποψη. Είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει κανείς να βάζει τρικλοποδιά στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά η οικονομική ανάπτυξη στην Ουγγαρία πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται ψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, 3%. Και μειώνεται και το δημόσιο χρέος. Οπότε, μιλάμε για οικονομικούς δείκτες της Ουγγαρίας που είναι θετικοί. Εμείς είχαμε μια οικονομία που ήταν σε, σε τραγική κατάσταση όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση. Η Ράτσο Καρθία ένα λεπτό. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ο Ισπανός Πρωθυπουργό είπε ότι θα είναι τα Χριστούγεννα της οικονομικής ανάκαμψης. Ο κύριος Βέμπερ είπε ότι οι χώρες όπου έγιναν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και στους δυο να πω ότι δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Τα λόγια τους είναι προσβολή για τις οικογένειες που χάνουν τις κατοικίες τους λόγω εξώσεων. Είναι προσβολή προς τους νέους που πρέπει να μεταναστεύσουν εκτός Ευρώπης για να βρουν δουλειά. Είναι προσβολή για τις οικογένειες και για τα άτομα που ε, έχουν ειδικές ανάγκες και που χάνουν τα δικαιώματά τους. Και τώρα προσπαθούν να αποδυναμώσουν και το φόρο επί των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό πνίγοντας τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη. Πρέπει να πληρώσουν αυτοί που φταίνε για αυτή την κρίση και από τους οποίους ποτέ δεν έχουμε απαιτήσει τίποτα. Μόνο έτσι μπορούμε να βγούμε από την κρίση με πιο δίκαιο τρόπο. Το οφείλουμε στους πολίτες μας. Όχι στους ψηφοφόρους, στους πολίτες μας. Ευζέντο Σενόφσκι Ένα λεπτό. Πρόεδρε, the eh, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με την Με συγχωρείτε, δεν έχουμε διερμηνία αυτή τη στιγμή. Να, επαληθεύσουμε αν γίνεται. Μπορείτε να ξαναρχίσετε. Pane dovolte mi stručně Πρόεδρε, επιτρέψτε μου πολύ γρήγορα να σχολιάσω το βασικό θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, είναι σαφές, ιδίως ε, στα δίκτυα, στις υποδομές, την καινοτομία και την έρευνα. Πρέπει όμως να διερωτηθούμε, διότι, γιατί οι ιδιώτες επενδυτές δεν είναι τόσο όσοι θα θέλαμε. Αυτά τα συζητήσαμε και στην περασμένη Σύνοδο Ολομέλειας. Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα του, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Αλλά έχω κάποιε ανησυχίε για του δύο πελίν, πυλώνε που έχουν προταθεί. 16 δι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 5 από την ΕΤΕ και καταλήγουμε στα 315. Γιατί Γιατί πρέπει να πάρουμε όμως κονδύλια όπως 3,5 δις από το από το CEF και από το Horizon 2020. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βιλίμσκι, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί εδώ δεν καταλαβαίνουν πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή μας. Έχουμε τρομερή ανεργία. Δεκαετίες είχαμε να έχουμε, να τόση ανεργία και τόση φτώχεια. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ανισχυτικά <clears throat> Και αυτό οφείλεται στην μεγάλη αστάθεια του ευρώ και στο γεγονός ότι με την πολιτική μηδενικών επιτοκίων αφαιρούμε ευημερία από την Ευρώπη. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πλειοψηφίας και του σώματος. Και μας λέγεται ότι θα υπάρξει επί 15 μόχλευση των ποσών που προσφέρονται και ότι αυτό θα μας φέρει ευημερία. Αυτά είναι αλχημία. Τι σημαίνει. Λένε ότι θα εξηγιανθεί η κατάσταση. Αλλά δεν είναι δυνατόν με αυτά τα μέσα να εξηγιανθεί. Κοιτάξτε, την εποχή των εθνικών νομισμάτων λειτουργούσε η Ευρώπη. Τώρα δεν λειτουργεί. Σας αφήνω να βγάλετε το συμπέρασμα ποια κατάσταση ήταν καλύτερα. Για οποιοδήποτε λογικό άνθρωπο είναι σαφέ. Ευχαριστώ. Δέχεστε την μπλε κάρτα του κύριου Λάιτφριντ, κύριε Βιλίνσκι. Κύριε Λάιτφριντ, 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, μα είπατε ότι είναι πολύ άσχημα τα πράγματα αλλά δεν μας λέτε τι πρέπει να γίνει. Δεν έχετε ιδέα για το τι να προτείνετε. Λέτε όχι, όχι, όχι. Λέτε ότι απλώς πρέπει ο καθένας να πάει στη γωνία του. Ο καθένας μόνος του έναντι των ε, τεράστιων πολυεθνικών επιχειρήσεων, των τεράστιων τραπεζών. Ξέρετε τι θα γίνει τότε. Τότε οι πλούσιοι θα γίνουν ακόμη ε, πλουσιότεροι και αυτοί οι οποίοι πρέπει να εργαστούν, τους οποίους εμείς εκπροσωπούμε, θα γίνουν ε, φτωχότεροι. Αυτό θα γίνει αν επιβληθούν οι ιδέες σας. Παρακαλώ κύριε Βιλίμσκι. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Α, ωραία. Κύριε Λάιφρεντ, αυτά που άκουσα είναι απλώς ε, προπαγάνδα. Πόσο λίγο λειτουργεί η κατάσταση είναι σαφές. Εδώ και δεκαετίες. Εδώ και δεκαετίες είχαμε εθνική, οικονομική και νομισματική πολιτική. Και παρόλα αυτά, τα κράτη-μέλη σε κάποιο επίπεδο φιλικά και ελεύθερα μπορούσαν να συνεργαστούν. Η πολιτική που προτείνεται τώρα εξυπηρετεί μόνο τις πολυεθνικές και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και το ξέρετε πάρα πολύ. Ξέρω ότι και σε διάφορους τομείς θα δώσετε περισσότερες δυνατότητε στους επιχειρηματικούς ομίλους και θα τους επιτρέψετε να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο σε ολόκληρη την Ήπειρό μας. Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής Πάουλου Ρανζέου. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Γιούνκερ, Πρόεδρε του Συμβουλίου. Σε πρώτη φάση ήθελα να εκφράσω την ε, εκτίμησή μου και την ικανοποίησή μου για την πρόταση επενδύσεων που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους μας. Απλώς θα πρέπει να, επιτρέψω την προσοχή σας στο εξή. Ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι αν δεν υπάρχει και μια διάσταση περιφερειακή, γιατί ασχολούμαι και με την πολιτική συνοχή, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε οι επενδύσεις να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των χωρών που μπόρεσαν να κάνουν τις απαραίτητες διευθυντικές μεταρρυθμίσεις. Οπότε η μόχλευση και η στήριξη για την αύξηση των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ώστε να υπάρξει επιτέλου και κοινωνική συνοχή. Και ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τι ε, προτεραιότητε τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα τη Ουκρανία και την ανησυχητική κατάσταση τη Ρωσία. Πέρα αμφιβολία μα ανησυχούν αυτά. Όμω κάτι που προέκυψε μόλι αυτή την εβδομάδα πολύ έντονα είναι το θέμα τη Τουρκία. Διότι βλέπουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε απλώ με την απειλή του Ισλαμικού κράτου, με τα προβλήματα στο βορρά με τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά μεταξύ των δύο τοποθετείται και η Τουρκία πλέον. Η Τουρκία με τα δικαιώματα και τα, τις βασικές ελευθερίες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα δώσω το λόγο σε, για μπλε κάρτα μόνο σε εκείνους που δεν είναι γραμμένοι στο κατάλογο μιλητών. Οπότε κύριε Ζωρίγκο δεν θα σας δώσω μπλε κάρτα, θα δώσω δυνατότητα έτσι και σε άλλους να πάρουν το λόγο. Επόμενος ομιλητής, Όλε λούτβιξον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ έχω τις αφιβολίες μου για το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί υπάρχουν πολλές υποσχέσεις, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, σύμφωνα με τα μαθηματικά πρότυπα τουλάχιστον, τα μοντέλα. Ναι, συμφωνώ με το γενικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε κύριε Γιούγκερ. Φυσικά πρέπει να κάνει επενδύσεις η Ευρώπη, είναι ζωτική σημασία και πρέπει να αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μας σήμερα. Είδαμε όμως ότι οι επενδύσεις ε, τώρα είναι 15% χαμηλότερες από ό,τι ήταν το 2007. Είναι σαφές επίσης ότι όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, αυτές οι επενδύσεις δεν θα αλλάξουν την κατάσταση, γιατί δεν αποτελεί πανάκια το επενδυτικό πρόγραμμα. Είναι βέβαια ένα στίχημα, είναι μια αρχή. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λύση, αλλά το ίδιο το πρόγραμμα δεν αποτελεί τη λύση. Ευχαριστώ, ήταν ακριβώς ένα λεπτό. Επόμενος ομιλητής, Μύροσλαβ Πιοτρκόφσκι. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, τα αποτελέσματα τη επόμενη συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υποτίθεται ότι θα εκφραστούν υπέρ τη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, σύμφωνα με τι ε, τελευταίε εκτιμήσει τη Eurostat, το ανακεφαλή ΑΕΠ δείχνει στρέβλωση τη οποιαδήποτε προσπάθεια οικονομική πρόοδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω η Ανατολική Ευρώπη, η Πολωνία, πλήττεται από την φτώχεια, όπω το Λούμπλιν, τα ανατολικά τη χώρα, με 44% σε σχέση με την Ευρωπαϊκή, υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ανακεφαλία ΕΠ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την εξωτερική μα βοήθεια και την πολιτική μα προ την Ουκρανία, όπω το χερσαίο δίκτυο συγκοινωνιών μας και την ε, μεταφορά, το μεταφορικό μας δίκτυο από την Βόρεια Θάλασσα, μέσω Λούμπλιν από την Βαρσοβία της Πολωνίας και ε, προς τα Βόρεια για να υπάρξει επικοινωνία με την Ουκρανία. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό η κυρία Λεπέν. Όταν ε, είμαστε μικρός πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη και όταν μεγαλώνουμε πιστεύουμε στο πρόγραμμα Juncker. 21 μικρά δισεκατομμύρια είναι γελίο να το συγκρίνουμε με τα 13-3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΤΕ. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία και κατά τη γνώμη σας θα έχουμε 294 από επενδύσεις. Πολύ ωραία. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθουν σε δημόσια σχέδια και προγράμματα τα χρήματα αυτά από τον ιδιωτικό τομέα, μάλλον επικοινωνιακό κόλπο είναι. Η πραγματικότητα είναι τα νούμερα και τα νούμερα της Ελλάδας για παράδειγμα που είναι στην επικαιρότητα. Εσείς εκεί στο βάθος που θέλετε να μας κάνετε μαθήματα. Η Ελλάδα λοιπόν, μείον Η ε, μειώθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, η λιγότερα νοσοκομεία, 35% ε, μειώθηκαν τα μέσα που δίνονται από 2007 μέχρι τώρα. 500 ευρώ είναι ο ελάχιστο μισθό και 300 για του κάτω από τα 25. 49,8% είναι οι άνεργοι κάτω των 25. 170% το χρέο Μπράβο. Συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα αυτά που έχετε στην Ελλάδα και οφείλονται στη δικιά σα οικονομική πολιτική. Υπάρχει μια μπλε καρτά από την κυρία Χάρμ. Τη δέχεστε? Με μεγάλη χαρά. Πιστεύετε ότι είναι σκόπιμη η επένδυση μετά αυτά που ακούσαμε χθε για τη Ρωσία. Θεωρεί ότι εφόσον ακούσαμε ότι η Ρωσία χθες έδωσε 40 εκατομμύρια σας έδωσε 40 εκατομμύρια για να καταπολεμήσει την Ευρώπη νομίζετε ότι αυτό είναι σκόπιμη επένδυση από πλευράς της Ρωσίας. Ως ήθιστε ό,τι να είναι, ό,τι περνάει από το μυαλό σα, Είναι ένα μακροχρόνιο σχέδιο. Αν δανείσαμε μια ρωσική τράπεζα, είναι γιατί μας ε, εμποδίζεται να χρηματοδοτηθούμε από τις γαλλικές τράπεζες και φταίει και το κόμμα σας που πολεμάτε όσους δεν είναι φίλοι σας. Το βασικό της πολιτικής σας είναι να βελτιώνετε την κατάσταση της οικονομικής αγοράς και των τραπεζών, ενώ εμείς θέλουμε να στηρίξουμε το λαό και όχι τις αγορές αυτές. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ότμαρ Κάρας, 1,5 λεπτό. Η πολιτική μας στοχεύει να ενισχύσει την ανεξαρτησία των κρατών μελών, τα, τη διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διατήρηση του εθνούς δικαίου και τη δημιουργία επενδύσεων, ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης, απασχόλησης. Κυρίες και κύριοι, ας έρθουμε τώρα στη συνάντηση κορυφής. Από αυτή τη συνάντηση κορυφής αναμένω να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι συγκεκριμένο και όχι απλώς να περασπίζονται την κατάστασή τους. Περιμένω τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν σοβαρά την πρόταση της Κομισιόν και να πάρουν αποφάσεις για εφαρμογή της αποφάσης αυτής και των αποφάσεων του Κοινοβουλίου. Περιμένω από τη συνάντηση κορυφής κάθε κράτος μέλος να συμβάλλει ούτως ώστε το πρόγραμμα Juncker για ανάπτυξη και απασχόληση να εφαρμοστεί συγκεκριμένα. Μπορούμε να διπλασιάσουμε τα 21 δισεκατομμύρια, να αυξήσουμε τις εγγυήσεις, να δώσουμε φορολογικά κίνητρα, μπορούμε να προτείνουμε προγράμματα. Προγράμματα. Προγράμματα ευρωπαϊκής προστιθέμενες αξίες και να μην περάσουμε σε επανεθνικοποίηση που να είναι βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά αντί να έχουν μεμονωμένα και παροδικά αποτελέσματα. Αυτό αναμένουμε. Σοβαρότητα και καμία εθνικοποίηση. Και προσβλέπουμε συγκεκριμένα να συνεχιστεί η δημοσιονομική εξυγίανση. Να συμβάλλουν σε αυτό όλα τα κράτη-μέλη. Να γίνουν πιο έντονες διαδοτικές μεταρρυθμίσεις για να υπάρχουν επενδύσεις. Και αυτό περιμένουμε από αυτήν τη συνάντηση κορυφή. Ευχαριστώ κύριε Κάρα. Ε, ο κύριο Χρυσόγονο θέλει να σα κάνει μια ερώτηση με μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Παρακαλώ. Μιλήσατε μόλι για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά η έκθεση σε σχέση με τα μνημονιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία συνυπογράφεται, διαπιστώνει ότι υπήρξαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια του ελληνικού προγράμματος και βέβαια δεν το διαπιστώνει μόνο η έκθεση το διαπιστώνουν και αποφάσεις παραδείγματος χάρη της επιτροπής του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη. ουσιαστικά με τα προγράμματα αυτά υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να παραβιάζουν υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. πώς το δικαιολογείτε εσείς αυτό; Κύριε Κάρας, 30 δευτερόλεπτα. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ήδη πριν από την ε, εκλογή του επανειλημμένα τόνισε ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έλεγχο της Τρόικα για αυτόν είναι σημαντικό στοιχείο για την μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε όλες αυτές οι παροδικές δομές που δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπίσουμε την κρίση να ξεπεραστούν και τότε θα μπορέσουν να εφαρμοστούν πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών. Και αυτή είναι η πολιτική μας. Ευχαριστώ κύριε Καράς. Ο κύριος ε, Ζουρίνιου για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, μετά τις ελπίδες που μας έφερε το πρόγραμμα της Επιτροπής Juncker, το πρόγραμμα εργασίας και τα συμπεράσματα που αναμένουμε από το Συμβούλιο είναι απογοητευτικά. Το μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξαρτάται από τα λόγια, εξαρτάται από τι πράξει. Οι Ευρωπαίοι και ο κόσμο θα κοιτάζουν τι συγκεκριμένε πρωτοβουλίε θα αναλυθούν. Και η διορία για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα είναι πολύ συγκεκριμένη. Το πρώτο εξάμεινο του 2015. Χάσαμε ήδη τι πρώτε μα ευκαιρίε και τώρα θέλουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων που να λειτουργήσει στην πράξη, να είναι χειροπιαστό, να, είναι απλώς, να μην είναι απλώ μια αποθήκη για προγράμματα που έμειναν στο χρονοτούλαπο και δεν βρήκαν καμία χρηματοδότηση. Να στηρίξουμε την Ενεργειακή Ένωση, να υπάρξει διαφάνεια και δημοσιονομική σύγκληση σαφή, αλλά και φορολογική. Να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία της ε, νομισματικής και τραπεζικής ένωσης. Πρόεδρε, η τελική, ε, αυτό που θα κρίνει το αποτέλεσμα θα είναι η δράση. Δράση ή απογοήτευση. Αυτό διακυβεύεται στο επόμενο Συμβούλιο. Και ήδη γνωρίζοντας τα συμπεράσματα όπως τα ακούσαμε σήμερα το πρωί, δεν έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κεφαλογιάννης. 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αν δει κανείς την πορεία των επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια εύκολα θα διαπιστώσει ότι από την παλιά ευρώπη των 10, των 15, των 28 κρατών έχει ουσιαστικά διπλασιαστεί. Όμως τώρα υπάρχει μια σημαντική υστέρηση 260 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακόμα και αν βγάλουμε, αν αφαιρέσουμε, αν εξαιρέσουμε τον τομέα των κατασκευών με την έκρηξή του στα τέλη της δεκαετίας του 2000 ε, θα διαπιστώσουμε ότι 160 δισεκατομμύρια γύπουν από το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πακέτο Juncker των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 16 δισεκατομμύρια του κοινοτικού προϋπολογισμού, τα 5 δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η μόχλεση των κονδυλίων, αλλά και η προσφορά, η συνεισφορά των κρατών μελών ασφαλώς και θα οδηγήσει και είναι η απάντηση στην κρίση επενδύσεων που έχουμε στην ευρωζώνη και στη δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας. Ο κύριος Γιούγκερ και ο αντιπρόεδρος του, ο κύριος Κατάινεν, έχουν πολύ σημαντική δουλειά να κάνουν. Πρέπει να ξεκινήσουν μια παγκόσμια εκστρατεία να πείσουν τους θεσμικούς επενδυτές, τις αγορές στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική, για να στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα των επενδύσεων το επενδυτικό ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι ένα στοίχημα που έχει θετικές αποδόσεις. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα στις αγορές. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να περάσουμε από την κουλτούρα των κονδυλίων του παρελθόντος στην κουλτούρα των επενδύσεων και της ανάληψης κινδύνων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Κεφαλογιάννη, δέχεστε μια μπλε του κυρίου Κύριε Φαρία, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν είναι ακριβώς για τον τελευταίο μας ομιλητή, για τον προηγούμενο ομιλητή ζήτησα τη γαλάζια κάρτα, αλλά τελικά δεν με δεχτήκατε. Θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, αλλά ε, μου ε, ανακοινώθηκε καθυστερημένα. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Κατλίν Φαν Μπρέμπτεν, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σας πω για ένα άνθρωπο που διάβασα στην εφημερίδα σήμερα που λέει ότι σπαταλάει σε αεροδρόμια η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα. Είναι επικεφαλή ενό άρθρου σε εφημερίδα. Και αναφήκε για την ε, Ισπανία, την Πολωνία, την Ελλάδα κλπ. Πάνω από 160 δισεκατομμύρια πηγαίνουν σε αεροδρόμια που φαίνεται ότι είναι χαμένα χρήματα. Γιατί δεν χρειάζονται τέτοιου είδου επενδύσει, γιατί δεν είναι αποδοτικά τα αεροδρόμια αυτά. Και βέβαια είναι πάντα πολύ ενοχλητικό για ανθρώπους που πιστεύουν στην Ευρώπη να διαβάζουν τέτοια άρθρα. Πρέπει να επενδύσουμε εκεί που πρέπει να επενδύσουμε. Και οι σοσιαλιστές και δημοκράτες Ξέρετε ότι θέλουμε πάρα πολύ να δώσουμε όθηση στο επενδυτικό αυτό πακέτο. Αλλά θέλουμε και μάλιστα ζητάμε από το Συμβούλιο να κάνει περισσότερα, να επενδύσει περισσότερα. Αλλά, αλλά όχι οπουδήποτε, όχι σε προγράμματα κύρους ή σε ένα ή άλλο κράτος μέλος, όχι, να επενδύσουμε στο μέλλον, με κριτήρια που να είναι το μέλλον, βιώσιμα προγράμματα που να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και αυτό το λέω και το τονίζω. Η ψηφιακή ατζέντα, για παράδειγμα, η κεφαλιακή ένωση, το περιβάλλον, αυτά είναι πράγματα για τα οποία χρειάζονται επενδύσεις, που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και όχι πράγματα τα οποία θα διαφημίσουν τους υπουργούς, πρωθυπουργούς της χώρες μέλη. Ο κύριος Κέλλη, μισή λεπτό τώρα. Δεν έχουμε και πολύ βεβαιότητα, αλλά έχουμε περισσότερη σαφήνεια για τις προθέσεις του κ. Γιούγκερ και για το επενδυτικό του πρόγραμμα. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε, διότι εάν ε, πετύχει, θα πετύχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αποτύχει, το ίδιο και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο έχει πολύ μεγάλες ευθύνες και το, Συμβούλιο θα πρέπει, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να το στηρίξει, όπως πάμε το πρωί. Από κάποιες οπτικές γωνίες ε, είδαμε ότι σωστά ο πρόεδρος Γιούγκερ ζήτησε από το Συμβούλιο να αναλάβει δέσμευση για αυτέ τι προτάσει και να δώσει τι απαραίτητε εγγυήσει για να προχωρήσουμε. Τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνε για να προχωρήσουν σε διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. Τι έχουν υποσχεθεί. Και όπω ο κύριο Βέμπερ είπε το πρωί, ε, είναι πολλά ε, τα. Είναι... Η Ιρλανδία που πριν από 4-5 χρόνια θεωρεί το μια αποτυχία, ε, έμαθε αυτά που έπρεπε να μάθει από την κρίση παρά το πόσο υπέφεραν οι πολίτε τη. Και φαίνοντα ει πέρα στι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κ. Γιούνκερ για την εμπιστοσύνη. Θα πει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε σχέσει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία. Ε, είναι πολλέ επιχειρήσει στην Ιρλανδία που ελπίζουν ότι του χρόνου θα μπορούσαν να προσλάβουν κι άλλων εργαζόμενο. Αυτό είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Διότι αν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση προσλάβει έναν ακόμη ε, εργαζόμενο, θα λύσουμε το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ευρώπη ή της οποιασδήποτε φούσκας απασχόλησης. Έτσι λοιπόν για την ανάπτυξη χρειάζεται η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και όχι το κενό. Ευχαριστούμε η κυρία Μίτση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Γιουνκέρ, κύριε Ντελαβεντοβά, η Ευρώπη πρέπει να ε, προχωρήσει και να αξιοποιήσει το οικονομικό της δυναμικό. Οι κοινωνικές εξελίξεις μετά την κρίση έδειξαν ότι δεν υπάρχει διάθε... Ε, τάση ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτό που τόσο καιρό λοιπόν αναμένουμε ε, είναι ακριβώς η στιγμή να κρίνουμε αν θα μπορέσουμε να το έχουμε με το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα. Εάν θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός, πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να ε, στηρίξουμε τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Ωστόσο, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες πρέπει να διευκρινιστούν από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πιο συγκεκριμένα, οι συνεισφορές των 100 μελών του ιδιωτικού τομέα τι ρόλο θα έχει, θα πρέπει αυτό να αποσαφινιστεί, καθώς και το πώς θα, ε, ποιος θα διευθύνει αυτό το ταμείο. Θα πρέπει να αποφύγουμε επίσης τη φοροδιαφυγή. Η επιτυχία του επενδυτικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την καλή οργάνωση. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητής είναι ο κύριος Χρυσιάνης Κάριν, 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Σήμερα μιλάμε για επενδύσει Τις χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Όμως πού θα βρούμε τις επενδύσεις αυτές. Ξέρουμε ότι το χρέος των χωρών μελών είναι τέτοιο που δεν υπάρχουν πόροι από εκεί. Οπότε από τον ιδιωτικό τομέα αυτό μας μένει. Ο ιδιωτικός τομέας έχει τα μέσα, παρόλα αυτά δεν επενδύει στην οικονομία. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν γιατί ο ιδιωτικός τομέας δεν επενδύει στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η απάντηση πιστεύω ότι είναι η εξής. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η ρύθμιση που ισχύει είναι πολύ ακαμπτή, πολύ βαριά. Δεν υπάρχει ευελιξία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα μας προτείνει μια λύση. Πώς θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε αυτές τις ιδιωτικές επενδύσεις για να πραγματοποιηθούν τα διάφορα προγράμματα. Με συνάδελφοι, αν οι χώρες μέλη δεν προχωρήσουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δεν θα έχουμε τις επενδύσεις αυτές από τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, πρέπει να βελτιώσουμε την ρύθμιση που είναι πολύ βαριά για τον ιδιωτικό τομέα και να ενισχύσουμε τα, τον προπολογισμό των χωρών μελών και να δαπανώνται τα χρήματα εκεί που πρέπει χωρίς πατάλες. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος λέει για ένα λεπτό. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι ξέρουμε την έκφραση ένας παππούς στο Skype στην Ουγγαρία διότι στην Ουγγαρία είναι πολλοί αυτοί που δεν έχουν την ευκαιρία, έτσι όπως είναι οργανωμένες οικογένειες, να συναντήσουν ε, τους παππούδες τους. Πολλές φορές πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη χώρα, γιατί εκεί είναι εγκατεστημένοι. Να λοιπόν, τι θέματα πρέπει να δούμε για χώρες που ε, στα ανατολικά της Ευρώπης έχουν μια πιο περίπλοκη κατάσταση. Στα ανατολικά της Ευρώπης δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί, δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικοί και 36.000 νέοι έφυγαν από την Ουγγαρία μόλις πέρσι. Δεν θα μπορούσε να έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε οι νέοι αυτοί να βρουν την θέση τους και όχι απλώς να μένουν σε επαφή μέσω Skype με τους παππούδες και τους γονείς τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. David Kaza. David Kaza 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Καταρχάς, Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Πρόεδρό της, τον κύριο Ζαν για αυτό το πολύ σημαντικό βήμα για την ε, περαιτέρω οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης. Κυρίως όμως θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Ένα άλλο θέμα που αντιμετωπίζει, την, ε, που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, το θέμα Ουκρανία-Ρωσία. την ε, προηγούμενη... Ε, συγγνώμη, θα μιλάμε για τα θέματα ε, αυτά, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα. Ε, υπάρχουν πολλά θέματα με τους πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται στην Μάλτα και η Μάλτα δεν μπορεί να παραμείνει μόνη για να αντιμετωπίζει τα κύματα των προσφύγων. Έχουμε πολλά κύματα προσφύγων, ιδιαίτερα από τη Βόρεια Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει κάνει πολλές προτάσεις και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη, το, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη-μέλη όμως ε, δεν μπορούν να καθυστερούν τόσο πολύ. Είναι κρίμα που η Ιταλική Προεδρία δεν αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Ενώ ε, τελειώνει η Προεδρία της. Δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζουμε έτσι τη χώρα μας. Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική αλληλεγγύη. Η Μεσόγειος έχει γίνει νεκροταφείο, είναι τρομερή ανθρώπινη τραγωδία δεν είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη να μην τρέπονται για αυτό που επιτρέπουν. Τώρα πρέπει να δράσουμε, όχι μόνο λόγια δράση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάζα. Και τώρα ο κύριος ε, Γκυγιόν Μπαλάς, ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ κύριε Γιούγκερ, κύριε εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Ακούσαμε τον κύριο Βέμπερ, τον κύριο Λάμπδορφ να λένε ότι η Γαλλία πρέπει να κάνει διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω να καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά παίζουν το παιχνίδι της κυρίας Λεπέν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θέλω να μιλήσω για την ουσία. Να θέσω το εξή ερώτημα. Υπάρχει μια τάση αποπληθωρισμού και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δεν υπάρχει βαθιά σχέση μεταξύ των διαθροτικών συναλλαγών, των φιλελεύθερων διαθροτικών ε, αλλαγών που θέλουν να μειώσουν και το εισόδημα και το κόστος εργασίας και αυτόν τον αποπληθωρισμό. Δεν υπάρχει σχέση σε αυτή τη στάση αναμονής που έχουν οι ιδιωτικοί επενδυτές εφόσον γνωρίζουν ότι γίνονται λίγες δημόσιες επενδύσεις και η αγορά είναι πεσμένη άρα οι επενδύσεις αυτές δεν καθησυχάζουν, δεν βοηθούν κανένα. Κύριε Γιούγκερ, δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο πρόγραμμα που παρουσιάζεται που λέει ότι οι δημόσιες πρέπει να είναι εγγύηση για τις ιδιωτικέ επενδύσεις και αυτή η κλίση για διαστοτικές μεταρρυθμίσει που δεν καθησυχάζει ούτε την αγορά ούτε του επενδυτές. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η επόμενη ομιλήτρια η κυρία Ελένη Θεοχάρους. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γιούνκε, εκπονήσατε φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη και είναι απαραίτητο να προχωρήσετε άμεσα και τάχιστα στην υλοποίησή τους γιατί οι λαοί της Ευρώπης και ειδικά οι φτωχοί λαοί του Νότου δεν αντέχουν άλλο. Οι οικονομίες των κρατών μελών είναι αλληλοεξαρτώμενες, ενώ σε ορισμένες χώρες που έχουν τεθεί σε σκληρά μνημόνια οι κοινωνίες είναι, εξακολουθούν να παραμένουν ταλαιπωρημένες, άστεγες, πεινασμένες ιδιωτικέ επενδύσει δεν μπορεί να γίνουν χωρί πολιτική και κοινωνική σταθερότητα και οι ανισότητε που υπάρχουν ω αποτέλεσμα τη απώλεια τη εργασία και των εισοδημάτων των πολιτών δημιουργούν σοβαρά πολιτικά προβλήματα τα οποία είναι εμφανή σήμερα στην Ελλάδα. Η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία αντιμετωπίζουν επίση σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Η ανεργία καλπάζει και η μετανάστευση είναι απειλητική ποιο θα επενδύσει σε συνθήκε πολιτική αστάθεια. η ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πολιτική κρίση και μερικοί επαναφέρουν το θέμα τη εξόδου τη από την ευρωζώνη με επιπτώσει σε όλε τι οικονομίε. αυτό αποτυπώνεται στα κρατικά ομόλογα και στα χρηματιστήρια πολύ σοβαρό αντίκτυπο θα υπάρξει και στην κύπρο που βρίσκεται επίση σε μνημόνιο και θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά. γι' αυτό θα πρέπει τώρα να στηριχθεί με κάθε μέσο η ελλάδα κύριε πρόεδρε. διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι θα προκληθεί συστημικό πρόβλημα που θα απειλήσει να τεινάξει το πρόγραμμα ανάπτυξη και την ευρωζώνη στον αέρα. σα ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι αποφασιστικό για να δούμε αν θα υπάρξει ανάκαμψη στην Ευρώπη. Η ομάδα των σοσιαλιστών είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Ιταλική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι χώρες μέλη θα σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους. Πρέπει να υπάρξουν λοιπόν δεσμεύσεις πρώτα για να υπάρχει ένα στρατηγικό ταμείο για επενδύσεις που είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε τι απαραίτητε στην Ευρώπη επενδύσει. Για να γίνει όμω κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν σε επίπεδο κεφαλαίου. Χρειαζόμαστε αυτέ τι εθνικέ συνεισφορέ να εξισορροπηθούν, να ουδετεροποιηθούν υπό την έποψη του Συμφώνου Σταθερότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η φορολογική πολιτική. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένα σημείο καμπή, όχι μονάχα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, αλλά και ώστε οι φόροι θα παραμένουν στις χώρες όπου προστίθεται αξία, όπου γίνεται η παραγωγή. Και αυτή ήταν η δέσμευση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτον, υπάρχει και η εντολή που δόθηκε στους τέσσερις Προέδρους για τη συμπλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Για να συμπληρώσουμε αυτή την Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε μια σύγκληση σε οικονομικό επίπεδο. Χωρίς τη σύγκληση η ευρωπαϊκή ζώνη, ευρώ, η ζώνη του ευρώ δεν έχει μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάιχτ Φρίντ για ένα μισή λεπτό. Schatten über Europa. Ein Schatten der Ungerechtigkeit. Das empfindet jeder. Jede Bürgerin, jeder Bürger ist unzufrieden mit dieser Ungerechtigkeit in der Europäischen Union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 ε, δεν ξέρω ελληνικά πώς γίνεται αυτό και βγαίνουν τα ελληνικά. Τώρα ακούγεται, τώρα είναι εντάξει. Μπορώ να μιλήσω ελληνικά, όχι, αγγλικά μπορώ να μιλήσω. Μπορείτε να συνεχίσετε. Όχι. Λοιπόν, αυτό και αν είναι άδικο, λοιπόν, αυτό και αν είναι άδικο. Υπάρχει μια αδικία στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το αλλάξουμε. Ε, συνοψίζω. Έχουμε φορολογική αδικία και αυτό θα πρέπει να ε, το ε, καταργήσουμε και θα πρέπει να υπάρχει και ισονομία και είναι μία από τις αξίες μας. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπορικές συμφωνίες όπου πηγαίνουν σε έκτακτα δικαστήρια ή μεγάλοι όμιλοι και ο μέσος πολίτης σε κανονικά δικαστήρια. Και αυτό αδικία είναι. Θα πρέπει να επανέλθει η δικαιοσύνη στην Ευρώπη που να είναι όλοι ίσοι και έτσι θα προχωρήσουμε στην Ευρώπη αλλιώς θα υπάρξει Σα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Μπορεί να μην με κατάλαβαν όλοι, επάντως συντήρησα το χρόνο μου. Ευχαριστώ πολύ και για την τήρηση του χρόνου. Παρά τα τεχνικά προβλήματα. Ο κύριος Τάνκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής ε, Juncker είναι μια καμπεί μια αλλαγή ε, νοοτροπίας περισσότερο στην πολιτική σκέψη παρά στην ε, οικονομία. Είναι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, βρεθούν κονδύλια και είναι μια πρόσκληση προς τα κράτη-μέλη και προς το Συμβούλιο να συνεχίσουμε να επενδύουμε. Αυτό που θέλουμε το του μελη δεν είναι λόγια να υποστηρίζουν τώρα το επενδυτικό σχέδιο, αλλά έργα. Να δημιουργήσουν εκείνο το οικονομικό πλαίσιο που θα βοηθήσει ε, να υλοποιηθεί αυτή η επένδυση. Και όσοι δεν το διαθέτουν να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις γιατί μόνο τότε θα δοθεί απαραίτητη όθηση για ε, ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Μόνο τότε θα δοθεί πραγματική όθηση και στους Ευρωπαίους και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κνούτ Φλέκενστάιν, τελευταίος ομιλητής για 1,5 λεπτό πριν από το ΚΑΤΣΙΑΙ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που μάθαμε από το, αλλά αυτά που περιμένουμε να μας πει το Συμβούλιο σε σχέση με την Ουκρανία. Περιμένουμε μία σαφή δήλωση και αποφασιστική δράση. Πρέπει να υπάρξει υποστήριξη για την νόμιμη κυβέρνηση της Ουκρανίας και για τον πρόεδρο Ποροσέγκο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη υποστήριξη για την εφαρμογή της ανακοχής που έχει συμφωνηθεί. Επομένως θα πρέπει να έχουμε σε επαφή και με τη Ρωσία. Πρέπει να δώσουμε υποστήριξη για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, ιδίως στην Ανατολική Ουκρανία. Υποστήριξη επίσης της εξέβρεσης μιας μορφής αποκέντρωσης και επίσης υποστήριξη για την υλοποίηση του σεβάθους, του προγράμματος σεβάθους μεταρρυθμίσεων που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει επομένως τίποτα ε, μέχρι στιγμή, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν οι άνθρωποι στην Ουκρανία ότι κάτι θα αλλάξει. Αυτό σημαίνει πραγματική πολιτική θέληση και οικονομική βοήθεια από τη δική μας πλευρά, ιδίως για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα κοινωνικά προβλήματα στη, στην φάση αυτή της μετάβασης που πρέπει να διαβεί η οικονομία της ε, Ουκρανίας και όχι μονάχα να δίνουμε λεφτά για τους προμηθευτές και τους εισαγωγείς. Μια μπλε κάρτα από τον κύριο Σούλτ. Θέλετε να τη δεχτείτε. Παρακαλώ. Με δίχως μικρόφωνο μιλτής Λέτε ότι ζητάτε οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία. Μα η Ουκρανία είναι ουσιαστικά χρεοκοπημένη. Και χρειάζεται δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ για να σταθεί στα πόδια της. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασώσει την Ουκρανία. Όπως έκανε με την Ελλάδα. Όχι ακριβώς διασώθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάστηκαν 250 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία πήγαν... Άρα, θέλετε να κάνουμε το ίδιο και με την Ουκρανία. 30 δευτερόλεπτα για την απάντησή σας. Αυτό δεν μπορεί να το πετύχει μόνο της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, χρειαζόμαστε οικονομική υποστήριξη για την Ουκρανία εάν θέλουμε να την διασώσουμε την Ουκρανία όπως είπατε μαζί με τα κράτη-μέλη, μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, μαζί με άλλους φορείς θα μπορέσουμε να το πετύχουμε και στο βαθμό που θα γίνουν και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία. Γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να δίνουμε λεφτά χωρίς να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη αλλαγή στην Ουκρανία. Και πιστεύω ότι όλοι μας το καταλαβαίνουμε αυτό και το υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Εννέα βουλευτές θέλουν επίσης να συμμετάσχουν στο Catch Eye. Σας παρακαλώ να παραμείνετε στο ένα λεπτό. Ε, Ματσάδες Πρέσο. Μεσέδες Μπρέσο μάλλον, συγγνώμη. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι μεταξύ των λίγων που θεωρούν ε, ότι το σχέδιο Juncker είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αν πραγματικά αποτελέσει το μέσο για να εισαχθεί ευελιξία για τα κράτη-μέλη, αλλά χρησιμοποιώντας τη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άρα με τρόπο που θα εγγυάται ότι όντως πρόκειται για επενδύσεις. Το ερώτημά μου αφορά και στρέφεται περισσότερο τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Προεδρίας δηλαδή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ότι δηλαδή τα κράτη μέσω επενδύσεων σχετικά περιορισμένων με τον μηχανισμό πολλαπλασιαστή επιταχυντή θα μπορέσουν να κάνουν πραγματικά αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη, δηλαδή να αυξηθούν εντόνως οι επενδύσεις. Επενδύσεις 300 δις, λέει το σχέδιο Γιούνκερ για τρία χρόνια, αλλά δεν αρκούν για να καλύψουν το κενό του ελλείμματος του επενδυτικού. Και αυτό μέσω της δέσμευσης όλων θα μπορέσει μόνο να λυθεί. Κύριος Μαριάς, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ε, Χθε αντί να κάνετε την αυτοκριτική σας για την παράνομη και ομή παρέμβασή σας στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας μου, υποστηρίξατε ότι στο όνομα της πολιτικής Ευρώπης και λόγω του ότι είναι γνωστή η πολιτική σας ταυτότητα, έχετε δίθεν το δικαίωμα να παρεμβαίνετε στα εσωτερικά της Ελλάδας σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι η συνθήκη της ευρωπαϊκής ένωσης επιβάλλει στην επιτροπή τήρηση πολιτικής ουδετερότητας. επιτέλους κύριε juncker σεβαστείτε τη συνθήκη της ευρωπαϊκής ένωσης και πάψτε να ενεργείτε ως εκπρόσωπο των δανειστών. σταματήστε κύριε juncker να ανακατεύεστε στα εσωτερικά της ελλάδας. ό,τι και να κάνετε κύριε juncker δεν μπορείτε να σώσετε τους μνημονιακούς πολιτικούς σας φίλους στην ελλάδα. η εκστρατεία κινδυνολογίας στην οποία έχετε επιδοθεί το τελευταίο διάστημα εσείς ο μοσχοβησίος σόιμπλε και η παρέα του δεν πρόκειται να περάσει. ο ελληνικός λαός στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα πετάξει έξω από την πατρίδα μας την τρόικα και τους ξένους δανειστές και θα προχωρήσει στη διαγραφή του του χρέους για τη δημιουργία του οποίου εσείς προσωπικά είστε υπεύθυνος. Ο το επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο οφείλει να πιέσει την τουρκία να πάψει να παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών όπω συμβαίνει σήμερα με την επίθεση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη κύπρου. πρέπει επίση να σταματήσει να καταπατεί τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα τόσο στο εσωτερικό τη με τη συλλήψη αντιπάλων τη και τη φήμωση του τύπου όσο και ενάντια άλλων κρατών. δυστυχώ ανταυτού ορισμένα κράτη μέλη προσπαθούν να προωθήσουν άνοιγμα κεφαλαίων της τουρκίας. το μόνο που μπορούν να επιτύχουν τέτοιες ενέργειες είναι να ενθαρρύνουν την τουρκία να συνεχίσει στην ίδια παράνομη και αντιδημοκρατική κατεύθυνση. αγαπητοί συνάδελφοι όσοι πραγματικά θέλουν να υπάρξει πρόοδο στην ενταξιακή πορεία της τουρκίας πρέπει να της υποδείξουν πως οφείλει να υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις να τερματίσει άμεσα τις απειλές και τις παράνομες ενέργειες να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συνεργαστεί για την επίλυση του Κυπριακού. Η κυρία Αναγκόμης έχει το λόγο. Ο δήμαρχος της Σύντρα της ε, πόλης από την οποία προέρχομαι είναι έτοιμος να ανοίξει σχολικά γεύματα όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους άνεργους εκεί. Δεν τρέπεστε κύριε Γιούνκερ που γίνεται αυτό σε μια χώρα την Πορτογαλία, που ορισμένοι όπως ο κύριος Βέμπερ πιστεύαν ότι θα γίνει η ατμομηχανή της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν χρήματα στο δημόσιο τομέα για επενδύσεις σε ανάπτυξη και σε απασχόληση, ενώ η φορολογική παράδειση στην Ευρώπη και αλλού συσσωρεύουν περισσότερα χρήματα και υπάρχουν και χώρες οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να μην πληρώνουν φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σκάνδαλο LuxLeaks έδειξε τις ευθύνες της Κομισιόν. Κάνουμε ένα αγώνα δρόμου προς τα κάτω, ένα φορολογικό dumping που καταπατά κάθε κανόνα φορολογικής εναρμόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν αδικία και εγκληματικότητα και διαφθορά η οποία περνάει μέσα από το δημοσιονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα εξωτερικά θέματα. Μην αφήσετε την κρίση στη Ρωσία, στην Ουκρανία και την Τουρκία να εμποδίζουν την απαραίτητη δράση σε επίπεδο Συμβουλίου για την διαμόρφωση μια πολιτική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να περιλαμβάνει και τη Λιβύη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρίνα Αλμπιόλ Γκουσμάν, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στο Ισπανικό κράτος γνωρίζουμε ήδη πάρα πολύ καλά τι εστί επενδυτικό σχέδιο Juncker. Δεν χρειάζεται να μας το εξηγήσει κανείς, γιατί ήδη ε, ε, το υφιστάμεθα ακόμα πριν εφαρμοστεί γιατί υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ήταν το πρόγραμμα Castor ε, για φυσικό αέριο στη θάλασσα με ομόλογα του Επενδυτικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 1,35 δις ευρώ στήχησε αυτό στον κρατικό κορβανά. 1,35 δις για τον κύριο Φλωρεντίνο Πέρες που είναι ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά κυρίως είναι πρόεδρος της τρίτης μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας του κόσμου. Ε, ε ο, ο ε, κρατικός εργολάβος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Αυτό είναι το πρόγραμμα ε, που επενεί μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άχρηστες. Αυτή είναι μια καλή περίληψη του ε, ε, σχεδίου Juncker. Πόσες επιταγές έχετε έτοιμες, σε ποια ονόματα. Για ένα λεπτό, επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Βάγκελ, εγώ κύριε Γιόνκερ θέλω να σας συγχαρώ για τις ε, φρέσκες ιδέες σας και για την ενέργειά σας. Ξέρω όμως πως ήδη έχετε κουραστεί σήμερα και θα είναι δύσκολο να μας ακούτε δύο μέρες. Ε, αλλά θέλω να εκφράσω μια επιθυμία εξ ονόματος των, των ε, ψηφοφόρων μας. Το επενδυτικό σας σχέδιο είναι καλό και το χαιρετίζουμε. Όμως οι ηλικιωμένοι ψηφοφόροι περιμένουν ένα σχέδιο το οποίο θα δώσει απαντήσεις και στις δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχετε θίξει και ελπίζω πως θα το πράξετε στις επόμενες σας παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γλέζος, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστό στην αρχή της ληστείας των λαών υπέρ του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα το οποίο όμως στηρίζεται και πάλι στη θεοποίηση του χρήματος. Δεν πρέπει να μας ξεγελάει το γεγονός ότι τα προτινόμενα μέτρα έχουν ντυθεί με τα κουστούμια της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα το Συμβούλιο μηχανεύεται με ποιο τρόπο θα προστατευθούν αντιλαϊκές κυβερνήσεις όπως στην Ελλάδα όπου ενώ η πραγματική δύναμη της κυβέρνησης υπολείπεται από το να έχει την πλειοψηφία έχει μόνο 106 έδρες χάρη στο καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα κλέβει 50 έδρες από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και αποκτά πλειοψηφία για να κυβερνά. Γι' αυτό ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού της Κομισιόν, ο Ζακ Γιούγκερ, επεμβαίνει με αντιδεοντολογικές δηλώσεις για να σώσει την οικία του κυβέρνηση. Δικαιολογήθηκε χθες ότι ως πολίτης έχει το δικαίωμα. Κύριε Γλέζο, να τελειώνετε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε γαλαζίες κάρτες στο ΚΑΤΣΙΑΙ. Δύο μιλητές ε, έχουμε ακόμα. Τη Βοσάνη και μετά η κυρία Φλασίκο Βαμπένοβα. Πρόεδρε, δύο πράγματα θα ήθελα να θίξω. Το ένα έχει ήδη αναφερθεί σε μια μπλε κάρτα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του κυρίου Γιούνκερ στο γεγονό ότι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αλλά και οι φορολογικέ απάτε δεν φταίνε για όλα τα προβλήματα που έχουμε με τους φόρους και με την εγκληματικότητα ε, όσον αφορά τους φόρους. Υπάρχει υπερβολική ε, ε, φορολογία και αυτό κάποιες φορές αναγκάζει την οικονομία να περάσει στην παραοικονομία. Ε, στην χώρα μου, την Ουγγαρία, έχουμε πολύ μαύρη αγορά λόγω του πολύ ψηλού ΦΠΑ. 27% είναι στα τρόφιμα και θα αυξηθεί κι άλλο από την κυβέρνηση. Οπότε αυτό αναγκάζει τους λιανοπολιτές των τροφίμων να περνά στην παραοικονομία. Ε, το άλλο θέμα είναι ότι το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να πάρει όλα τα ποσά από τα υπάρχοντα ποσά. Κυρία Μπένοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γιούνκερ, θα έχετε να αντιμετωπίσετε πάρα πολλά προβλήματα τις επόμενες μέρες. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει βελτιωθεί από μόνη της. Αυτό κοστίζει πάρα πολύ στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του εμβάρδου. Αυτά τα χρήματα λοιπόν τα χρειαζόμαστε για την οικονομία μας, για τον εαυτό μας. Ένα άλλο ζήτημα <clears throat> όπου τα πράγματα επιδεινώνονται συνέχεια είναι η οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μου έχει φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο η αμοιβή των εργαζομένων. Είναι πάρα πολύ υψηλή η ανεργία. Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν ένα πρόβλημα το οποίο θα λύσετε εσείς και πρέπει το Συμβούλιο Κορυφής να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτόν τον χρόνο που έχουμε ενώπιόν μας ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, δουνε να βρουν μια λύση στα προβλήματά τους. Ο κύριος Γιούνκερ λοιπόν θα λάβει τώρα το λόγο. Σας παρακαλώ να παραμείνετε μόνο στα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, θαυμάζω την εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ που έχετε. Ε, αλλά δεν πειράζει, ας είναι και αστεία αυτή η έκκληση και η παράκληση. Κανονικά θα έπρεπε να φύγω στις 10 και μισή. Αλλά κάθισα μέχρι το πικρό τέλος και ε, πρέπει να απαντήσω σε ένα λεπτό. Έχουν γίνει ερωτήσεις εχθές, προχτές, έχουν απαντηθεί αυτές σε προηγούμενες συζητήσεις. Γιατί ε, πρέπει να είμαι υποχρεωμένος να ξανααπαντήσω. Και στο μεταξύ πολλοί ε, ε, από αυτούς που έκαναν ερώτηση έχουν αποχωρήσει από την ολομέλεια Θα ήθελα να επαναλάβω για να είναι σαφές. Για το επενδυτικό αυτό σχέδιο, για να μπορέσουμε να το ε, εφαρμόσουμε, χρειαζόμαστε επιγόντως τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ε, τα αντίστοιχα κείμενα που θα σας έρθουν τον Ιανουάριο και ελπίζω το Κοινοβούλιο ε, να αντιδράσει γρήγορα. Και χρειάζεται και δραστήρια αντιμετώπιση και υιοθέτηση από τις κυβερνήσεις. Καλό είναι να διαβάζει εφημερίδες κανείς, ε, τις οποίες διαβάζω κι εγώ, αλλά όχι αρκετά συχνά. Και έχω μάθει ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον έξι ε, πρωθυπουργοί είπαν ότι καλό το κοινοβούλιο, έχουν γίνει πρώτα ε, βήματα, αλλά είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Μέχρι σήμερα κανείς δεν είπε πόσα δισεκατομμύρια θέλει να συνεισφέρει για τις εγγυήσεις και θεωρώ ότι αύριο και μεθαύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κατακλειστεί ε, από προσφορές των τραπεζών. Να δούμε το τι έχει υποθεί τις τελευταίες εβδομάδες σημαίνει ότι θα θησαυρίσουμε και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να ε, αυξηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Ε, το επενδυτικό σχέδιο εκείνη από κάποια κρατικά κονδύλια όπου μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να αυξηθούν ε, τα χρέη και χωρίς να υπάρξουν προβλήματα για τους προϋπολογισμούς. Άρα θα πρέπει να κινητοποιηθούν χρήματα και από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για τις επενδύσεις και στην πραγματική οικονομία μάλιστα. Και ποιο ε, θα επενδύσει στην Ευρώπη δηλαδή αν δεν είναι αυτό το ιδιωτικό κεφάλαιο που έχει πάρα πολλά χρήματα. Ναι, ναι. Δηλαδή πάλι ο φορολογούμενος θα την πληρώσει αντί να την πληρώσουν αυτοί που έχουν αρκετά χρήματα. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί και συνοδεύει αυτά τα προγράμματα, αλλά δεν τα υλοποιεί η ίδια. Το επαναλαμβάνω. Όταν το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον καλείται πολύ να το πράξει. Γιατί να το κάνει η Επιτροπή. Υπάρχουν εμπειρογνώμονε που ξέρουν την οικονομία, που είναι της αγοράς. Ε, θα πρέπει να αναβάλουν, ε, συγγνώμη, να αναλάβουν αυτή την ευθύνη, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί θα αρχίσουν να γκρινιάζουν κυβερνήσει και ευρωβουλευτές. Ότι καθυστερούμε, ότι ολιγορούμε, ότι δεν υλοποιούμε τα προγράμματα. Υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να υποστηριχθούν, που μακροπρόθεσμα έχουν δυνατότητα ανάπτυξης. Δεν θέλουμε να χτίσουμε νέες, ε, ε, νέους καθεδρικούς ναούς. Έχουμε ένα σωρό παρεκκλήσια και εκκλησάκια. Ε, ε, δεν θέλουμε έργα βιτρίνας. Θέλουμε έργα για τα έργα και όχι έργα για τα μάτια. Και θα πρέπει να ε, διασκεδάσουμε και αυτή την εντύπωση ότι δεν έχουμε υπόψη μας ε, τίποτα κοινόνα ε, θεωρητικά, ότι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε, λέει, κάποια πυρηνικά εργοστάσια και την πυρηνική ενέργεια. Καμία σχέση. Το ενεργειακό μείγμα είναι και παραμένει εθνική υπόθεση και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά, κυρία Πρόεδρε, στα γαλλικά τώρα, δεν με εντυπωσιάζουν καθόλου εκείνοι που εδώ και λίγες μέρες με καλούν να μην ε, λέω τίποτα και κάποιοι άλλοι μου λένε να μιλώ. Γιατί ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι άραγε ο μόνο που δεν έχει το δικαίωμα να λέει τη γνώμη του και να εξηγεί τι πεπιθήσει του. Εδώ συζητάτε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ συχνά μάλλον, ε, όχι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ως Εθνικά Κοινοβούλια που αντιπαρατίθενται. Εγώ πολιτικός είμαι και μην ε, προσπαθείτε να με ε, φημώσετε. Θα έχω ε, και θα λέω ό,τι θέλω να πω. Αν αφορά αυτό μια χώρα θα το λέω. Όλος ο κόσμος μπορεί να επικρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σιωπά. Ε, λοιπόν δεν πρόκειται να σιωπήσει. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Και εγώ σας είχα δώσει ήδη λίγο χρόνο παραπάνω. Δεν χρειάζεται να διαμαρτύρεστε. <coughs> και τώρα εξ ονόματος του Συμβουλίου, ο κύριος Πενεδέτο Ντελαβέντοβα, έχει το λόγο όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λιγότερο από πέντε λεφτά εγώ θα μιλήσω. Αξιότιμοι συνάδελφοι, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Εγώ παραμένω στα όσα ήδη ανέφερε η Κομισιόν. Εγώ δεν μπορώ να προτρέξω των αυριανών ε, πορισμάτων του Συμβουλίου. Πάντως, ε, τις ε, παραγωγικές, στην παραγωγική, πλαίσιο παραγωγικής συνεργασίας θα διαβιβάσω τις προσδοκίες, τις παρατηρήσεις, τις επικρίσεις, αλλά και την ενθάρρυνση που προέκυψε γενικώ, αλλά και το τομεακώς όσον αφορά την συζήτηση που αφορά το επενδυτικό σχέδιο, το σχέδιο Juncker όπως ε, καθιερώθηκε να λέγεται. Αυτό το Συμβούλιο θα είναι το πρώτο υπό την ε, ε, ηγεσία του νέου Προέδρου Ντόναλτ Τούσκ και του νέου Προέδρου της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Αν και οι δύο είναι νέοι στα αξιώματά τους, έχουν ε, μακρά πείρα που έχει αποκτηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπως, ορισμένα από, όπως και ορισμένα από τα μέλη του Κοινοβουλίου εξάλλου. Επειδή ε, κλείνει και η Ιταλική Προεδρία, θα ήθελα να τους ευχηθώ τις καλύτερες με ευχές όχι μόνο για το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ επικοδομητικό, αλλά και για το μέλλον και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση.